Okay, um, good morning everybody. I've waited. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, περίμενα λίγο. Ε, καθυστέρησα λίγο την έναρξη, περιμένω τους συναδέλφους. Πάντως με ιδιαίτερα χαρά θα ήθελα να καλωσορίσω τον Μπέρναρτ Χόιερ, που είναι πρόεδρος, Ευρωπαϊκής, ε, που είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι η μεγαλύτερη ε, δημόσια Τράπεδα επενδύσεων στον κόσμο και ε, είναι ενδιαφέρον να δούμε ποιοι ενδιαφέρονται εδώ για επενδύσεις στην Επιτροπή μας. Εγώ σίγουρα ενδιαφέρομαι πάρα πολύ και ο Βέρνερ θα μας παρουσιάσει το έργο της ΕΤΕ και φυσικά θα ακολουθήσει ένας γύρος ή περισσότεροι έρωτα απαντήσεων. Βέρνερ. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, είναι λίγο δύσκολο μετά από 25 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνηθίσω στην ιδέα ότι δεν είμαι πια ευρωβουλευτής, αλλά το πνεύμα το έχω κρατήσει ακόμη. Ευχαριστώ, αισθάνομαι μεγάλη χαρά για την πρόσκληση, τιμή ιδιαίτερη, αλλά και υποχρέωση, γιατί όπως είπατε κι εσείς, η ΕΤΕ είναι η μεγαλύτερη τράπεζα, δημόσια τράπεζα επενδύσεων και μάλιστα είναι και μοναδική στη φύση και το χαρακτήρα της, γιατί είναι πλήρως υπόλογη στα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Γιατί η ΕΤΕ ιδρύθηκε με βάση τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τις διαπραγματεύσεις της συνθήκης της Ρώμης. Οπότε η ιστορία της ΕΤΕ συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά. Και φυσικά οι επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μια πολύ τιμητική και φυσικά απαραίτητη λειτουργία της ΕΤΕ. Γι' αυτό και είμαι στη διάθεσή σας και ελπίζω να σας φανεί χρήσιμη αυτή η συζήτηση. Η ΕΤΕ είναι τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Η μέτοχή της δηλαδή, είναι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν δώσει μια σαφέστατη εντολή, δηλαδή να συμβάλλουμε στους στόχους και στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Και βάση αυτού του επιχειρησιακού μοντέλου της ΕΤΕ είναι οι εγγυήσει των μετόχων της τράπεζας καθώς και η επιμονή σε ένα χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας, κάτι που επιτρέπει στην τράπεζα να συγκεντρώνει κεφάλαια στις ε, χρηματαγορές και να το μεταβιβάζει με πολύ ευνοϊκά επιτόκια. Είναι σημαντικό λοιπόν να το αντιληφθούμε αυτό. Δηλαδή, η δέσμευση των κρατών μελών φυσικά είναι ευπρόσδεκτη για μας και απολύτως απαραίτητη ε, και αυτό θα το αναφέρω μετά ως προς την ε, αύξηση του κεφαλαίου αλλά στόχος της τράπεζας είναι να πηγαίνει στις ε, χρηματαγορές και να δανείζεται από τις κεφαλαγορές, από τις χρηματαγορές σε ευνοϊκά επιτόκια λόγω της θέσης και μετά αυτό το χρηματοπιστωτικό πλεονέκτημα να το μετακυλεί στους υπόλοιπους ε, παραλήπτες. Και είναι κάπως δύσκολο αυτό, αυτή, ε, ότι αποτινόμαστε στις χρηματαγορές. Γι' αυτό και το προσέχουμε ιδιαίτερα. Θα είμαι σύντομος σε ό,τι αφορά το δεύτερο σημείο, την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το 2011. Έχει περάσει αρκετός καιρό. Όλα τα θετικά στοιχεία της έκθεσης δεν έχουν μία σχέση με μένα, γιατί εγώ ανέλαβα τέλος, τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου αν γίνουν καλά το 2012 θα ευθύνομαι εγώ, αλλά για το 2011 με φόρο τιμή στους προκατόχους. Πέρυσι ήταν μια χρονιά τεράστιων προσπαθειών, εργοδόν προσπαθειών για την τράπεζα. Μετά την κατάσταση της Lehman Brothers το 2008 και την κρίση και μας ζητήθηκε από τους μετοχές να αυξήσουμε τις δανειστικές μας δραστηριότητες για να ξεπεράσουμε την κρίση και τότε σκεφτήκαμε να ε, μετά από δύο χρόνια να, εμφανιστούμε σε επίπεδα, ε, να επανέλθουμε σε επίπεδα πριν τη ε, κρίση, ελπίζοντα ότι η κρίση θα περνούσε γρήγορα. Η διεύρυνση των χρηματοδοτικών μα και των δανειστικών μα δραστηριοτήτων σημαίνει περισσότερα δάνεια. Και το 2011 πήραμε 76 δισεκατομμύρια από τι διεθνεί χρηματαγορέ. Δανειστήκαμε 76 δισεκατομμύρια. Έτσι μπορέσαμε να χρηματοδοτήσουμε 400 54 σχέδια σε 70 χώρες. Με βάση το επιχειρησιακό μας σχέδιο επενδύσαμε κυρίως σε οικονομία της γνώσης, σε προγράμματα δράσης για την ενέργεια και το περιβάλλον, σε δίκτυα μεταφορών, σε 74 οργανισμούς που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περίπου 100.000 ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με βάση την εντολή μας, και διαπίστωσε ότι έχετε ζωηρό ενδιαφέρον γι' αυτό, 10% των δραστηριοτήτων μας ε, κατευθύνθηκαν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν των δανειστικών μας ε, δραστηριοτήτων, ένα άλλο σημείο είναι η παροχή συμβουλών και ε, φυσικά δανεισμός, συνεργασία, συμβουλή. Φυσικά ο δανεισμός είναι αυτονόητη δραστηριότητα μιας τράπεζας. Το blending το 2011 συνδυάσαμε ε, πόρους ε, της κοινότητας των κρατών μελών και της ΕΤΕ για διάφορους μηχανισμούς επιμερισμού κινδύνου και οικονομικό προγραμματισμό. Και ως εκ τούτου είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων προς την Επιτροπή σας για την ε, εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και φυσικά είμαι ευγνώμων και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί στήριξε αυτή τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΕΤΕ. Σε ό,τι αφορά την παροχή συμβουλών ε, και ως προς αυτές τις συμβουλευτικές δραστηριότητες, έχουμε πολύ περισσότερους μηχανικούς ε, εμπειρογνώμονες και επιστήμονες στην τράπεζα από ότι τραπεζίτες. Η παροχή τεχνικών συμβουλών ε, προς τους πελάτες μας αυξήθηκε αισθητά όχι μόνο λόγω της κρίσης του χρέους στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, το 2011 είναι πίσω μας πια. Γι' αυτό και θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τις μελλοντικές προκλήσεις της τράπεζας. Όταν οι μέτοχοί μας αποφάσισαν ότι η τράπεζα θα πρέπει να διευρύνει τις δραστηριότητες της ε, αισθητά μάλιστα μετά το 2008 και μετά να κατεβεί σε επίπεδα πριν την κρίση. Δεν σκέφτηκαν οι μετοχοί ότι μετά από αυτό θα μας χτυπούσε και η κρίση χρέους δεν το είχαν προβλέψει. Μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση είχαμε και την κρίση του δημόσιου χρέους που συνεχίζεται και σήμερα. Γι' αυτό και το σχέδιο επαναφοράς σε επίπεδα πριν την κρίση, μετά τα πρώτα χρόνια, μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, γιατί σε τελική ανάλυση, με μια τέτοια προσπάθεια και ουσιαστικά φέτος αυτή την πορεία ακολουθήσαμε να επιστρέψουμε σε τέτοια επίπεδα, δρούμε με τρόπο αντισυγκυριακό, αντικυκλικό και ε, αντιβαίνει στα, στα μακροοικονομικά μας ένστικτα και στις μακροοικονομικές μας τάσεις. Αν θέλουμε ε, να μιλήσουμε τώρα, να δράσουμε αντικυκλικά και όχι προκυκλικά, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στους περιορισμούς. Και ο περιορισμό είναι η επαναφορά σε επίπεδα 2008-2009, ακόμη και 2011 θα ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Οπότε τα εξηγήσαμε όλα αυτά στα κράτη-μέλη. Και είναι κάτι πολύ δύσκολο σε μια εποχή όπου όλοι πασχίζουν να αντιμετωπίσουν την κρίση χρέους στη χώρα τους και την δημοσιονομική κρίση μάλλον. Και αν εμείς θα διευρύνουμε και πάλι της, το δανεισμό μας. Αυτό θα πρέπει να γίνει με μια πιο εύρωστη κεφαλαϊκή βάση. Το κεφάλαιο της τράπεζας είναι 232 δισεκατομμύρια. Τεράστιο ποσό, υπέρογκο. Δυστυχώς όμως, τα κράτη-μέλη αποφάσισαν πριν από δεκαετίες να χρηματοδοτούν μόνο, να καταβάλουν μόνο το 5% αυτού του κεφαλαίου. Οπότε έχουμε 11 δις από τα κράτη-μέλη. Επιπλέον έχουμε τα κέρδη των δεκαετιών που δεν μοιράστηκαν ε, ως μερίσμα των συμμετόχους, έμειναν στην τράπεζα και αυτό είναι περίπου 50 δις. Ο συνολικός μας δανεισμός όμως είναι δεκαπλάσιος από αυτά τα ποσά. Οπότε ήταν σαφές ότι έχουμε εξαντλήσει τα όρια των ε, κανονιστικών ε, λόγων που πρέπει να τηρήσουμε. Γι' αυτό εξηγήσαμε στα κράτη-μέλη ότι μία αύξηση του όγκου του δανεισμού θα σήμαινε ή θα, θα, θα προϋπέθεται μία ενίσχυση του κεφαλαίου, του pay-in κεφαλαίου, του κεφαλαίου που συνέβαλαν εισέφεραν τα κράτη-μέλη. Και ε, προς μεγάλη έκπληξή μας συμφώνησαν τα κράτη-μέλη. Δεν έχει γίνει ακόμη βέβαια. Συμφώνησαν επί χάρτου. Θα πρέπει να ληφθεί και η επίσημη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των ε, των κυβερνητών, των διοικητών. Πάντως, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου συμφώνησε για μια αύξηση του κεφαλαίου της ΕΤΕ. Είμαι πεπισμένος ότι είναι μια πολύ ισχυρή δέσμευση, στεναρή δέσμευση των κρατών μελών απέναντι στην τράπεζά μας και θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε το όγκο δανεισμού την επόμενη τριετία κατά 20 περίπου δισεκατομμύρια το χρόνο. Κάτι που δεν θα είναι εύκολο. Μην, Μην πιστεύετε ότι σε κάθε γωνία μας περιμένουν τα τέλεια σχέδια και προγράμματα. Η τράπεζα θα πρέπει να επιμείνει σε χρηματοδότηση υγιών, καλών, πολλά προγραμμάτων. Και γι' αυτό ζήτησα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας υποστηρίξει για τον προγραμματισμό αυτών των σχεδίων. Πρέπει, θα έπρεπε να αναμειχθούμε και στην διαμόρφωση ε, στην ανάπτυξη και δρομολόγηση των προγραμμάτων και σχεδίων ε, σε προγενέστερο στάδιο. Γιατί υπάρχουν πολύ καλοπροαίρετοι ε, στην άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν πολύ καλές ιδέες, τις δημοσιεύουν μάλιστα μερικές φορές και έχουν μεγάλη απήχηση στην κοινή γνώμη. Αλλά όταν φτάνουμε στο τεστ, στη δοκιμή, στη λιδία αλήθεια της οικονομικής βιωσιμότητας του προγράμματος, τότε η τράπεζα λέει όχι. Και αυτό είναι κίνδυνος για την ε, φήμη. Εδώ θα πρέπει να εμπλέκονται όλοι. Γι' αυτό και θα πρέπει η ΕΤΕ να συμμετέχει στη διαδικασία από τα προκαταρκτικά στάδια. Για να φαίνεται από την αρχή και να διαγνώσουμε από την αρχή αν είναι βιώσιμο οικονομικά το, το α ή β σχέδιο ή όχι. Τα κράτη-μέλη γνωρίζουν ότι θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους επιπλέον μας στόχους όχι μόνο για την Ευρωζώνη, αλλά για τα 27 και σύντομα και 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο όμως εφόσον η τράπεζά μας θα παραμείνει σε μια ισχυρή θέση ε, δανειστή στην αγορά και δανειζόμενο φυσικά. Γιατί είμαστε και μεγαλύτερη, είμαστε μεν η μεγαλύτερη δημόσια ε, τράπεζα επενδύσεων, αλλά είμαστε και ο μεγαλύτερος ε, δανειζόμενος θα πρέπει να συνεχίσουμε να μπορούμε να δανειζόμαστε με ευνοϊκά επιτόκια και να μπορούμε να χρηματοδοτούμε καλά προγράμματα και να κρατήσουμε την καλή μα θέση στην αγορά. Α μην το ξεχνούμε αυτό. Και <laughs> το 3α, αυτό είναι εν συντομία η έκφραση της καλή θέση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα τρία γραμματάκια τα 3α, είναι η έκφραση τη εμπιστοσύνη τη αγορά. Ε, ε, για αυτό που κάνουμε. 76 δισεκατομμύρια πήραμε φέτος από τις ε, διεθνείς αγορές και τα μισά ήταν από μη ευρωπαϊκές πηγές. Θα πρέπει λοιπόν να το κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας. Γιατί μιλούμε για έλλειψη αξιοπιστίας και εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Αλλά περίπου 40 εκατομμύρια εμείς τα πήραμε εκτός της Ευρωπαϊκής Ευρώπης. Αυτό σημαίνει πόση εμπιστοσύνη έχουν οι εξωκοινωτικοί δανειστές στην Ευρώπη. Α μην μιλούμε λοιπόν για έλλειψη εμπιστοσύνη. Επίση, μερικέ φορές μας κατηγορούν για υπερβολική επιφυλακτικότητα, για αποφυγή κινδύνου, κινδυνοφοβία. Λάθος. Μία τράπεζα αναλαμβάνει κινδύνους, αλλά πρώτα απ' όλα διαχειρίζεται του κινδύνους και νομίζω ότι το κάνουμε με αρκετή σύνεση. Η διαφύλαξη λοιπόν του τριπλού α δεν είναι αυτός σκοπό. δεν είναι θέμα εικόνα. Είναι θέμα οικονομικής πραγματικότητας, σκληρής οικονομικής πραγματικότητας. Αν δεν κρατήσουμε αυτή την θετική αξιολόγηση, δεν θα μπορούσαμε και εμείς να μετακυλήσουμε στους τελικούς παραλήπτες μας αυτό το θετικό αποτέλεσμα της εικόνας μας και της θέσης μας. Γιατί και έτσι θα πλήξουμε και τις χώρες που έχουν καλές δραστηριότητες και δανείζονται με χαμηλά επιτόκια. Και εμείς ε, ανταγωνιζόμαστε με αυτές την αγορά, οπότε θα μπορούσε κανείς να πει γιατί να, γιατί να εξακολουθούμε να είμαστε στις όχι για να παραγωνίζουμε άλλους, όχι για να ε, εξωθούμε άλλους εκτός της αγοράς ή να πλήξουμε τον ιδιωτικό τομέα. Και από τη στιγμή του χαρτοφυλακίου, από την άψη του χαρτοφυλακίου της τράπεζας, και της ευρωστίας του χαρτοφυλακίου της τράπεζας, είναι σημαντικό να έχουμε δάνεια και προς χώρες που είναι σε καλή κατάσταση. Είναι εύρωσης. Γι' αυτό και λέμε ότι η τράπεζα θα πρέπει να είναι παρούσα σε όλα τα κράτη-μέλη και με προγράμματα και φυσικά με τις δανειοληπτικές της δραστηριότητες. Τώρα είμαι στη διάθεσή σας να μιλήσουμε για τους διάφορους μηχανισμούς που έχει αναπτύξει η Τράπεζα και η Επιτροπή. Ήταν πραγματικά μια επιτυχία από το RSFF στο RSI, τα γνωρίζετε όλα αυτά. Έχουμε και ε, με την πρωτοβουλία για τα project bonds, για τα ομόλογα έργου. Έχουμε ένα νέο εργαλείο στην εργαλειοθήκη μας. Περιμένουμε τον Οκτώβριο την ε, υπογραφή την επίσημη και εκεί θα διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο. Και αυτό είναι ένα επιπλέον εργαλείο στην εργαλειοθήκη μας. Δεν είναι και καμία πανάκια. Θα πρέπει να δούμε ποιε θα είναι οι πρώτε μα εμπειρίε από αυτό το θέμα, γιατί θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η απόφαση για την επιτυχία του PVI θα εξαρτηθεί από την κατεύθυνση των αγορών. Γι' αυτό και είναι σοφό, συνετό και σκόπιμο η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να σκεφτούν όχι με τα πιο δύσκολα σχέδια στην πιλωτική φάση, αλλά τα πιο υποσχόμενα, πιο πολλά υποσχόμενα πιο πιθανά να σημειώσουν επιτυχία για να δώσουν μεγαλύτερη όθηση σε αυτό το νέο εργαλείο. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι έχω θέσει τις αδερές γραμμές και ένα πλαίσιο στο, και στο μέλλον θα επιτύχουμε σε αυτή την ε, ακροβασία μεταξύ του να είμαστε ένα υπεύθυνο θεσμικό όργανο, υπόλογο απέναντι στα κοινωτικά θεσμικά όργανα και αφετέρου και μια τράπεζα με ένα συντηρητικό ρόλο. Και με ιδιαίτερη χαρά θα έρχομαι να σας ενημερώνω και να συζητώ μαζί σας τις δραστηριότητες τράπεζας, όποτε το κρίνετε χρήσιμο. Σας ευχαριστώ. Uh, thank you very much. Um... Σας ευχαριστώ. Έχουμε τώρα κοινή συζήτηση των σημείων 13 και 14 της ημερήσιας διάταξης. Το 14 αφορά τη δική μας έκθεση επί της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Οπότε θα έχουμε κοινή συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και ερωτήσεις. Μια και έχουμε τη χαρά της παρουσίας του Προέδρου της ΕΤΕ, του Βέρνερ Χόιερ. Θα δώσω λοιπόν το λόγο τώρα στο Μάριο Μάουρο, που είναι ο εισηγητής της έκθεσης για να πει μερικά λόγια, ίσως να θέσει ερωτήσεις. Μετά θα ακούσουμε τους σκιώδη εισηγητέ ή οποιοδήποτε άλλο θέλει να λάβει το λόγο. Λάγκε, Γκίγκολτ, Γκίλαρ, Βολφ Κλίντς, ο Νικόλας Χουντής που είναι και σκιώδης, Θεόδωρος. Yeah, Dirk, you're a shadow, so you're all... Dirk, όλοι έχουν περιληφθεί στον κατάλογο. Θα ακούμε δύο-τρεις συναδέλφους και αν ε, θέλετε κύριε Χόιερ να απαντήσετε μπορείτε να μου κάνετε νόημα. Ο Μάριο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μου φάνηκε να κατάλαβα ότι έχω το χρόνο για να παρουσιάσω σύντομα το περιεχόμενο της έκθεσής μου. Πρώτα απ' όλα όμως, θα ήθελα πριν από την παρουσίαση να κάνω την απευθείας μια ερώτηση στον Πρόεδρο και αυτό και παράλληλα και με τις προτεραιότητες που έθεσα στην έκθεσή μου. Είναι πολύ απλή η ερώτησή μου. Εσείς παραδειγματικά μας παρουσιάσατε πόσο αυξήθηκε ο στρατηγικός ρόλος της ΕΤΕ. Εγώ ρωτώ και με την συνεισφορά όλων των συναδέλφων πώς η έκθεσή μου μπορεί να χρησιμεύσει για την υποβολή προτάσεων, όχι απλώς για μία περίληψη των πρεπραγμένων. Και η ερώτηση δεδομένης της αλλαγής σεναρίου, δεδομένου και του ρόλου της τράπεζας που κατάφερε να πείσει τους μετόχους για αύξηση του κεφαλαίου, εσείς θεωρείτε ότι χρειάζεστε ένα θεσμικό upgrade, μια θεσμική αναβάθμιση. Θέλετε μία αλλαγή του καταστατικού λειτουργίας της ΕΤΕ, ώστε να είστε ελεύθεροι να πράξετε εκτός ε, φυσικά από όλα εκείνα τα κεφάλαια που αφορούν τη διαφάνεια της τράπεζας. Θεωρείτε δηλαδή κύριε Πρόεδρε ότι το θεσμικό προφίλ της ΕΤΕ θα πρέπει ή θα μπορούσε να τύχει βελτιώσεων ούτω ώστε να παίξει μεγαλύτερο πρωταγωνιστικό ρόλο στο σενάριο της οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας τα ρωτώ αυτά, διότι θα ήθελα η έκθεση για την οποία συζητάμε να μην επικεντρωθεί μόνο στην, στην κριτική του, των περισσινών πεπραγμένων αλλά σε προτάσεις οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες για την μελλοντική δραστηριότητα. Εσείς αναφέρατε και εγώ εξάλλου το αναφέρω η αύξηση του τριπλού αλφα και η αύξηση του κεφαλαίου είναι στοιχεία κλειδί. Και αυτό μας επιτρέπει με μια σχετική ασφάλεια να αναλάβουμε την πιλωτική φάση των project bonds και που για μένα θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα στο τέλος του 2013. Ένα άλλο σημείο που θέλω να ληφθεί απόψη, υπόψη είναι μια πιο άμεση ε, εμπλοκή της ΕΤΕ στην, στα ευρωπαϊκά σχέδια, σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, φυσικά πάντοτε παραμένοντας το ρόλο της. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ορισμένες προτεραιότητες παρέμβασης υποδιερώντας τις ιεραρχικά. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή μέσα στην Ένωση και έξω από την Ένωση. Ελπίζω και να με ενθαρρύνουν και όλα οι συνάδελφοι να συνεχίσουμε να επικεντρώνουμε την προσοχή μας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναπτύσσοντας όμως περαιτέρω και τα ε, μέσα για την μικροοικονομία όπως και την οικονομική, κοινωνική οικονομία ενισχύοντας τα δίκτυα μέσα στις περιφέρειες διότι το πλαίσιο το, μέσα στο οποίο κινείται η ΕΤΕ είναι ένα πλαίσιο 500 εκατομμυρίων ανθρώπων και 23.000 ΜΜΕ και αποτελούν το 8% της, ε, του, του, παγκόσμιου πληθυσμού αλλά κατέχουν το 58% του welfare, του παγκοσμίου welfare, της παγκόσμιας ευημερίας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε μία εναλλακτική λύση για να διαφυλάξουμε αυτό το welfare που με σας εσείς είπατε ότι έχει πεθάνει λόγω της συγκυρίας. Επίσης, προτεραιότητες σε διεθνές πλαίσιο. Εσείς θυμήσατε και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στις επενδύσεις στις χώρες της Μεσογείου και να κρατήσουμε τις υποσχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αραβική Άνοιξη και τις δηλώσεις της Δοβίλ του 2008. Η ΕΤΕ επένδυσε στον τομέα των υποδομών, ΜΜΕ και συνέβαλε στις οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις επιτόπου. Τελευταίο, ρωτώ διαφάνεια και έλεγχο. Πολλές φορές ζητήθηκε από την ΕΤΕ να ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο και κυρίως τις χρηματοδοτήσεις που έχει δώσει με διαμεσολαβητές, με μεσάζοντες σε τρίτες χώρες. Εμείς ε, σήμερα που μιλάμε για τραπεζική εποπτεία, κατά τη γνώμη σας, τι σχέση θα πρέπει να θεσπίσουμε μεταξύ ΕΤΕ και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κατά τη γνώμη σας η ΕΤ θα πρέπει να ε, υπόκειται στον έλεγχο της ε, Κεντρικής Τράπεζας, αυτό υπό τη λογική της τραπεζικής εποπτείας. Ο κύριος Ευχαριστώ. Καταρχάς καλώς όριστε στην Επιτροπή μας. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, είχα κάποιο πρόβλημα με το αυτοκίνητο, αλλά έφτασα. Θα ήθελα να θίξω ορισμένα ζητήματα τα οποία πάντα, στα οποία πάντα αναφέρομαι όταν ε, γίνεται λόγος για την ε, ΕΤΕ. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και είναι και ο ρόλος μας εξάλλου να αναφέρουμε συνέχεια αυτό το πρόγραμμα έτσι ώστε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων και να έχουμε δημιουργική και η συζήτηση. Μέσα στα πλαίσια της κρίσης η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων νομίζω πως παίζει πολύ σημαντικό ρόλο παρέχοντας ανάπτυξη στην πραγματική οικονομία. Και αυτό πιστεύω ότι είναι και ο κύριος στόχος της έτσι κι αλλιώς. Ε, με τα λύπης είδα πως η κρίση του 2008 έφερε τα επέδα της οικονομίας χαμηλότερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και το συνολικό κεφάλαιο θα έπρεπε να δοθεί σε επενδύσεις. Αυτό θα ήταν κάτι καλό. Γι' αυτό πρέπει να ζητήσουμε αύξηση του επενδυτικού κεφαλαίου για τα επόμενα χρόνια. Επίσης, με τα χαράς ε, είδα ότι η πιλωτική περίοδος εγκρίθηκε και σχετικά με αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τον ε, Πρόεδρο ποιο είναι το ε, καθεστώς τώρα του project τι γίνεται. Κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικά προβλήματα όσον αφορά τους μεσάζοντες και τους δικαιούχους. Λίγα πράγματα γίνονται, δημοσιοποιούνται στο κοινό και οι περιοριστικές δυνατότητες, ε, είναι κάτι στο οποίο χρειάζεται να επενδύσουμε έτσι ώστε να προστατευτούν οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Κάτι άλλο, σημαντικό εξίσου, είναι οι φορολογικές οάσεις. Κάτι που δεν έχει επιληθεί ακόμα. Η πολιτική της τράπεζας στο ζήτημα αυτό είναι ανεπαρκής, διότι δεν διασφαλίζει δημόσιο χρήμα στην ευρωπαϊκή πολιτική, χρησιμοποιείται για άλλες περιπτώσεις. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από την ε, ΕΤΕ να αυτοαξιολογηθεί να διεξάγει τη δική της αξιολόγηση. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, οι πρόσφατες ε, εξε... Ε, τι γίνεται με τις πρόσφατες εκθέσεις για τους φορολογικούς παραδείσους. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι ανυπομονώ για μια στενή συνεργασία με τον κύριο Μάουρο και με τους υπόλοιπους σκιώδεις εισηγητές σε αυτό το φάκελο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Θεόδωρος Κυλάκης. Ε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χόιερ, για την παρουσίασή σας. Είπατε ότι με το νέο πακέτο θα διαθέσετε 60 δισεκατομμύρια στα επόμενα τρία χρόνια. Θα μπορέσετε να αυξήσετε τον, ε, τις πιστώσεις. Τι γίνεται όμως με τα υπόλοιπα 40 δισεκατομμύρια του ε, συνολικού πακέτου των 100 δισεκατομμυρίων για την αύξηση κεφαλαίου. Τι γίνεται με αυτά. Θα διατεθούν ας πούμε στα επόμενα 2-3 χρόνια μετά. Και πώς αναμένεται ότι θα είναι τα επιτόκια δανεισμού ε, στα επίπεδα που είναι τώρα ή αναμένεται ότι θα αυξηθούν. Και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είπατε ότι υπάρχουν 27 κράτη-μέλη. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη στα οποία τα επίπεδα ανεργίας είναι τρομακτικά υψηλά. Και πιστεύω ότι τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια θα έχουν ένα τέταρτο του πληθυσμού τους άνεργο. Εσείς πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε τη διαφορά όσον αφορά τα επίπεδα ανεργίας. Πιστεύετε ότι οι επενδύσεις αυτές μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά ή η διαφορά στα παιδανεργία θα είναι οριακή. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αναφέρθηκαν πάρα πολλά ζητήματα και ο Βέρνερ δεν έχει χώρο πια να τα σημειώσει. Γι' αυτό ακόμα βέβαια έχουμε να τον ρωτήσουμε πολλά, αλλά ας του δώσουμε χρόνο να απαντήσει το πρώτο σκέλος των ερωτήσεών σας. Αν τα καταφέρετε Βέρνερ, πέντε σε πέντε λεπτά. Δύσκολο. Θα προσπαθήσω πάντως. Ευχαριστώ. Καταρχήν κύριε Μάουρο, θερμά ευχαριστώ για το εξαιρετικό έργο σας και την προσπάθεια και τη δική σας και των συναδέλφων σας στα πλαίσια της έκθεσής σας και ευχαριστώ που θέσατε και κάποιες ερωτήσεις για το μέλλον γιατί Καλό είναι να κοιτάμε και να εξετάζουμε και το παρελθόν. Αλλά το Φεβρουάριο είχα παρουσιάσει την έκθεση του 2011. Έρθει η ώρα λοιπόν να ταινίζουμε και το μέλλον και να μην κοιτάμε μόνο προ το παρελθόν. Στρατηγικό ρόλο τη ΕΤΕ. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπω είπα, ιδρύθηκε ε, στο πλαίσιο τη συνθήκη τη Ρώμη. Και αυτό φαίνεται. Γιατί η διακυβέρνηση, η, της τράπεζας είχε αποφασιστεί τότε από τη συνθήκη της Ρώμης. Και τότε η οικονομική κοινότητα παρτίζονταν από έξι μέλη. Φαντάζεστε λοιπόν πως κάθονταν και κανόνιζαν το καταστατικό για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τότε είχαν στο μυαλό τους ένα επιπλέον master plan, Marshall, ε, σχέδιο Marshall, ιδιαίτερα για την Ιταλία τότε. Ε, μέχρι και σήμερα το γραφείο μας στη Ρώμη είναι το μεγαλύτερο γραφείο. Και αυτή ήταν η ιδέα. Ναι. Μην επαναλάβουμε το σχέδιο Marshall στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, αλλά να το επικεντρώσουμε εκεί που θα ήταν πιο απαραίτητο. Και η διακυβέρνηση της Τράπεζας δεν, είχε δεν ήταν προετοιμασμένη για μια Ευρώπη που θα παρτίζεται από 27 μέλη. Οι δομές της Τράπεζας, λοιπόν, είναι τέτοιες που κάποιοι ε, όπως είχαν επινοήσει κάποιοι στο, στον Περσί και στη Βόνη το 1956. Θα πρέπει να το σκεφτούμε λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, ε, έχει εργαστεί σωστά. Ήταν κρυμμένη στα δάση του Λουξεμβούργου αρχικά και έχει μετατραπεί στη, στο μεγαλύτερη ε, τράπεζα του κόσμου δι, δι, επενδύσεων και ε, μεγαλύτερο δανειολήπτη έχει τεράστια επίπτωση και στα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα θα πρέπει να ξεφύγουμε, να βγούμε έξω από τα δάση του Λουξεμβούργου και να διαδραματίσουμε το ρόλο μας με διαφάνεια, με άνοιγμα και σε στενή σχέση και συνεργασία με τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και ιδιαίτερα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει γίνει μεγάλη πρόοδος διανοητική ε, όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί είπαμε θα πρέπει να αναμίξουμε το βασικό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη του Κοινοβουλίου με τις ε, ε, δανειοδοτικές δραστηριότητες της τράπεζας. Αυτό είναι το θέμα, να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Γιατί είναι πολύ ωραία αυτά που λέμε και συνθήκες του ανταγωνισμού, είναι πολύ δημοφιλή και φυσικά και εμένα με ενδιαφέρει ο ανταγωνισμός ε, και δεν απορρίπτω τις συνθήκες, ε, τις συνθήκες ανταγωνισμού. Το αντίθετο. Και είμαστε ε, υπόλογοι και στο ελεκτικό συνέδριο και σε εσά και δεν έχουμε ε, μη Ευρωπαίους ε, μετόχους σε ισχυρές θέσεις τράπεζες. Είναι μια πραγματικά δηλαδή ευρωπαϊκή τράπεζα αυτή. Να το έχετε υπόψη. Έχετε μια τράπεζα που είναι αποκλειστικά ευρωπαϊκή. Και εκεί πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο της τράπεζας. Ο ρόλος της τράπεζας είναι, όσο πιο ισχυρός είναι και όσο πιο σαφής και διαφανής είναι, θα πρέπει ε, φυσικά και να μπορεί να πει όχι σε ένα σχέδιο. Και θα πρέπει να μπορούμε να λέμε ε, στις χώρες μέλη, ωραίο πρόγραμμα, αλλά δεν ε, είναι βιώσιμο. Να μην μας ε, πιέζουν να χρηματοδοτήσουμε σχέδια που δεν έχουν ε, νόημα από οικονομική άποψη. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Γιατί το τριπλό α, όπως σας είπα, δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά είναι ανάγκη. Και αν έχετε ε, ε, επίγνωση ότι ε, μερικοί μέτοχοι μόνο στα όνειρά τους βλέπουν πια το τριπλό α από εμά. Εμείς έχουμε καταφέρει και το διατηρήσαμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη θέση μας. Και οι χρηματαγορές, οι κεφαλαγορές εντυπωσιάστηκαν που οι μέτοχοι ενέκριναν την αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας που ελπίζουμε τελικά θα δεθεί σε εφαρμογή. Άμεση ανάμειξη της ε, τράπεζας ε, σε τραπεζικές ε, ικανότητες και φυσικά χαιρόμαστε για την σχετική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικεντρωθούμε. Θα συνεχιστεί η έμφαση που δίνουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 120.000 είχαμε πέρυσι και σε μερικές ειδικά χώρες μέλη και του ευρώ και εκτός της ευρωζώνης, οι δραστηριότητες των εμπορικών τραπεζών μειώνονται δραστικά. Και θα επιδεινωθεί η κατάσταση και με τη Βασιλεία 3. Οπότε πρέπει να καλύψουμε ένα κενό, εμείς οι ΕΤΕ, για να μην ε, πληγούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πήγα την περασμένη εβδομάδα, κύριε Σκυλακάκη, στην Αθήνα για να συνάψω συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση με αποκλειστικό στόχο τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και θέλουμε να το αναπτύξουμε αυτό το σχέδιο. Ο κύριο Λατσαρόλη ε, διαπραγματεύθηκε το πακέτο αυτό με την Ελλάδα και θα το αναπτύξουμε περαιτέρω γιατί το πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μερικέ φορέ ε, δεν φαίνεται εκ πρώτη όψεω. Μιλάμε για εργαλεία τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης και πρόβλημα η Ελλάδα έχει μερικές φορές με την εισαγωγή εγγύσεων, γιατί έχουμε επιτυχημένε αγωγών, γιατί έχουμε επιτυχημένες ε, επιχειρήσεις ε, ε, στην διεθνή αγορά, αλλά δεν μπορούν να, κάνουν τις εισαγωγές που χρειάζονται στην εταιρεία τους. Τέτοιου, τέτοια εργαλεία και μηχανισμούς προσπαθούμε να αναπτύξουμε. Σε ό,τι αφορά τα επιδόκια δανεισμού, αν μπορούσα να προβλέψω τι ύψο θα έχουν, θα ήμουν πανευτυχή. Πάντω η παρούσα κατάσταση είναι μάλλον καθησυχαστική. Έχουμε πραγματικά εκτόνωση στην αγορά μετά την απόφαση της ΕΚΤ πριν από δύο εβδομάδες. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε πια να αναπνεύσουμε. Α, συγγνώμη, να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου σας. Θα επιταχύνω. Δύο λόγια για τη διαφάνεια και την ε, λογοδοσία. Σε ό,τι αφορά την συμμόρφωση, εμείς θέλουμε να είμαστε καλύτεροι. Γι' αυτό και ενισχύσαμε τη θέση μας και εντός της τράπεζας και εκτός, ώστε για θέματα φορολογικών παραδείσων λοιπά είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και προσεκτικοί. Τώρα, για τη Μεσόγειο και τον ε, υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε συγκεκριμένη εντολή από το Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαίρομαι για αυτή για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους της Ένωσης. Και αυτό που κάνουμε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποβαίνει εις βάρος των δραστηριοτήτων μας εντός της Ένωσης. Γιατί η ιδίαυλη χρηματοδότηση είναι διαφορετική και η Μεσόγειος είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα. Αν ε, έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες ανταπεξέλθει πραγματικά στις υποχρεώσεις τους που απέρευσαν από την Αραβική Άνοιξη. Αφιβάλλω. Η τράπεζα κάνει ό,τι μπορεί. Καλή συνεργασία με την BERT και την Παγκόσμια Τράπεζα. Και έχουμε πολύ έντονες δραστηριότητες εκεί. Και παρόλο που είχαμε δυσκολίες με, ε, με τις ε, πρεσβείες που κάηκαν την περασμένη εβδομάδα, πάντως στη Λευκοσία είχαμε συνάντηση αποφασίσαμε τελικά να χρηματοδοτήσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα υποδομών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για, τη βορεια, για τις βορειοαφρικανικές χώρες. Ευχαριστώ. Πάντως είστε, μπορείτε να είστε βέβαιοι θα απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις, αν όχι σήμερα, σίγουρα γραπτός. Νομίζω το πρόβλημα της ανταλλαγής απόψεων είναι ο χρόνος, οι ερωτήσεις και απαντήσεις και των σχεδόν εισηγητών και όλων. Αυτό που νομίζω ότι θα κάνω είναι πριν επανέλθω, θα λάβω όλες τις ερωτήσεις ε, από την Επιτροπή γραπτά, γιατί χρειαζόμαστε και κάποιο χρόνο να τις επεξεργαστούμε και θα επανέλθω σε εσά, διότι δυστυχώς πρέπει να τελειώσουμε στην ώρα μας. Εάν υπάρξει λοιπόν πίεση χρόνου, θα δώσω προτεραιότητα σε εκείνους που διατύπωσαν τις ερωτήσεις τους εδώ. Ε, συμφω... Ε, Σβέν, θα το κάνεις εσύ, αν δεν κάνω λάθος. Θα μιλήσω γερμανικά. μια και έχουμε Γερμανό πρόεδρο. Λοιπόν, έχω ορισμένε ερωτήσεις που θα ήθελα να διατυπώσω και θα σας παρακαλούσα αν θέλετε να, το κάνετε, να τις διατυπώσετε γραπτές τις ερωτήσεις να τις κάνετε. Αλλά καταρχάς, Ευρωπαϊκός, έχουμε έναν ξεκάθαρο στόχο το 2015 να προχωρήσουμε με τον οδικό χάρτη για μια ε, καινοτόμο οικονομία, αλλά φτωχή σε διοξίδιο του άνθρακα, σε εκπομπή, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Τι γίνεται με τις επενδύσεις στα εργοστάσια παραγωγής ε, ενέργειας που χρησιμοποιούν ε, άνθρακα. Ο στόχος είναι να μειωθούν οι εκπομπές κατά 80 ή 95%. Εμένα θα με ενδιαφέρε να μάθω Τι γίνεται με την ε, στρατηγική, πόσο σοβαρά έχετε πάρει τη στρατηγική, πόσο την αντιμετωπίζετε, πόσο... Πού, πού έχει φτάσει η στρατηγική για τις ε, μειώσεις. Ιδιαίτερα όσον αφορά την περίπτωση της Γκλένκο, η ΜΚΟ για πολλούς μήνες έπρεπε να ασκήσουν πίεση στην τράπεζα, έτσι ώστε η τράπεζα να πάρει στα σοβαρά το έργο της και χαίρομαι που το αποτέλεσμα ήταν καλό. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τι αποκομίσατε από αυτό τι και πώς θα το χρησιμοποιήσετε σε άλλα project, ε, εάν η τράπεζα προτίθεται να τηρήσει τις υποσχέσεις της, ασκώντας πίεση σε άλλες επιχειρήσεις ε, οι οποίες ε, χρήζουν αξιολόγησης. Επίσης, ποιες είναι οι επιπτώσεις από την περίπτωση Γκλένκο. Επίσης, κάτι άλλο. Τον τελευταίο χρόνο δημιουργήθηκε μια ιδιαίτερη συμφωνία με την ΕΚΤ, έτσι ώστε η πρόσβαση στις ε, προδιαγραφές ρευστότητα να βοηθήσουν την ε, τράπεζα, διότι η τράπεζα μπορεί, θα τα χρειαστεί αυτά. Αναρωτιέμαι όμως, εάν είναι αναγκαία αυτή η συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, διότι η ΕΤΕ έχει στη διάθεσή της το, τον, ε, τον ESM, το ESFF, Αλλά χρειάζεται και η σύμφωνη γνώμη ώστε να υπάρξει πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια. Και η διαφάνεια είναι ένα ζήτημα που χρήζει συζήτηση και θα ήθελα διευκρινίσω όσον αφορά τη διαφάνεια του πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Προς το παρόν αυτά, ξανά ευχαριστώ και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το έργο σας. Και πραγματικά ανησυχώ όταν υπάρχει τόση μεγάλη πίεση και πολιτική πίεση για το έργο της ε, ΕΤΕ, ε, γιατί τότε πραγματικά θα χρειαστείτε την βοήθειά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, επόμενος και ο εισηγητής. Ο κύριος Χουντής. Οπότε παρακαλώ θερμά να μην ξεπεράσετε το τρίλεπτο για να προλάβουμε να μιλήσουμε όλοι. Είναι δίκαιο για όλους πιστεύω κάτι τέτοιο. Ε, Νικό, ε, κύριε Χουντή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θα το ξεπεράσω το τρίλεπτο διότι ε, θέλω να καλωσορίσω και εγώ τον Πρόεδρο της Τράπεζας Επενδύσεων ε, να μου επιτρέψει να κάνω ορισμένες ερωτήσεις που έχουν σχέση με αυτό που ανέφερε και αυτός πριν Δηλαδή πριν μια εβδομάδα ο κύριος Πρόεδρος επισκέφθηκε τη χώρα μου, την Ελλάδα, και όπως μάθαμε υπεγράφει μια συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση για χρηματοδότηση υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η είδηση αυτή πήρε μεγάλη δημοσιότητα και ήταν δημοφιλής για τους λόγους που όλοι γνωρίζετε. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω κύριε Πρόεδρε είναι επειδή αυτή την είδηση ότι θα υπάρξει βοήθεια της Τράπεζας Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Την έχουμε ακούσει στην Ελλάδα δύο φορές και μάλιστα ε, αυτή τη χρονιά, δηλαδή το 2012. Δηλαδή χρονιά που είστε, αν κατάλαβα καλά και σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο, πρόεδρος. Μπορείτε να μου πείτε λοιπόν τι εγγυάται ότι αυτή τη φορά θα γίνουν πραγματικότητα αυτές οι συμφωνίες, αυτές οι υποσχέσεις με την εγγύηση της τράπεζάς σας θα χρηματοδοτηθεί η δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Τι ήταν εκείνο που το εμπόδιζε μέχρι τα τώρα, ενώ είχε εξαγγελθεί δύο φορές. Αυτό θα με βοηθήσει να καταλάβω και ε, ε, την ευρύτερη πολιτική και στρατηγική που ακολουθεί η τράπεζά σας. Και το δεύτερο, από την επίσκεψή σας κύριε Πρόεδρε βγήκε μια ανακοίνωση στην οποία ε, λέτε τη συμφωνίας με την ελληνική κυβέρνηση ότι αυτή η συμφωνία που υπογράψαμε ανοίγει το δρόμο για την εκταμείευση δανείων για έργα όπου προαπαιτούμενο είναι η εγγύηση της ελληνικής δημοκρατίας. Εδώ αντιλαμβάνεστε, το ερώτημα είναι τι εννοείται εγγύηση της ελληνικής δημοκρατίας. Δηλαδή μέχρι τα τώρα ή υπάρχει θέμα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα ελληνικά ομόλογα και μια δεύτερη και τελειώνω πλευρά, ποια έργα αν έχετε υπόψη σας, θα χρηματοδοτηθούν μέσω αυτής της συμφωνίας. Το μόνο που ξέρουμε εκεί είναι οδικά έργα που έχουν σταματήσει διότι οι τράπεζες δεν, δεν έχουν παράσχει μέχρι τα τώρα τις ε, απαραίτητες εγγυήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις εφόσον είσαστε πρόχειρος. Είναι πάρα πολύ σημαντικές και για μια άμεση ενημέρωση αλλά και για να μπορέσω να έχω μια καλύτερη εικόνα για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η τράπεζά σας. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Τέκ, ε, για την ομάδα ICR. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εκ μέρους της ομάδας μου, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χόιρ για την παρουσίασή του και να αναφέρω περιληπτικά πώς βλέπουμε εμείς το ρόλο της ε, ΕΤΕ καλούμε την ε, τράπεζα να συνεχίσει τις καλές τραπεζικές πρακτικές και να διατηρήσει μια ισχυρή θέση όσον αφορά το κεφάλαιο σε μια φιλελεύθερη αγορά. Ε, φυσικά καλωσορίζουμε τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων, διότι πιστεύουμε ότι η ΕΤΕ ε, μπορεί να γίνει ακόμα πιο διαφανής όσον αφορά τις δανειστικές επιχειρήσεις της, ιδιαίτερα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα θέλαμε να μάθουμε τις απόψεις σας προς το παρόν όσον αφορά τα ομόλογα έργου για την Ευρώπη 2020, ιδιαίτερα όσον αφορά την, ε, την, τον καταμερισμό του κινδύνου και την τιμολόγηση. Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω για την δυνατότητα απορρόφησης ε, χωρών της Μεσογειακής Ευρώπης. Ελπίζουμε η οικονομική ανάπτυξη να επανέλθει αλλά εσείς πώς βλέπετε τη δυνατότητα απορρόφησης εκεί, διότι σε πολλές περιπτώσεις χώρες όπως για παράδειγμα η Ισπανία έχουν αεροδρόμια, σιδηροδρομικό δίκτυο, δικό δίκτυο, πώς εσείς μπορείτε να επενδύσετε έτσι ώστε να προωθήσετε την ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Διότι αυτό είναι καθοριστική σημασία, η επαναφορά τη ανάπτυξη δηλαδή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα προχωρήσαμε, εκτός από τους κοιότητες συζητητές, τους επόμενους ομιλητές. Πρώτος ο κύριος Βέρνερ Λάνια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μας παρουσιάσατε την ετήσια έκθεση του προκατόχου σας. Δεν την διάβασα όλη, είναι αλήθεια. Αλλά είδα ότι από τα 4.635 project 590 είναι στην Ισπανία, 700 περίπου στην Ισπανία, 146 στην Ελλάδα. Αυτά έχουν εφαρμοστεί. Ε, ρωτώ, πώς αξιολογείτε εσείς ως ΕΤΕ την ε, δυνατότητα στην Ευρωζώνη να εφαρμοστούν περισσότερα ε, έργα που προωθούν την ανάπτυξη. Και η δεύτερη ερώτηση που ήθελα να κάνω είναι όσον αφορά τα πιλωτικά έργα τα επιλοτικά ομόλογα έργου, με συγχωρείτε. Είπατε ότι τον Οκτώβριο θα ληφθεί απόφαση για τον ε, όγκο. Ε, μας αναφέρατε 32 εκατομμύρια για όλα αυτά τα project συνολικά. Αναφέρθηκε η πίεση από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πίεση που θα μπορούσε να είναι τόσο μεγάλη έτσι ώστε να επηρεαστεί η ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων της ΕΤΕ. Επίσης, άλλη ερώτηση όσον αφορά τους ε, τομείς του οποίους διαμοιράζονται τα έργα αυτά που έχετε εκρίνει στην Ευρώπη των 27, πιστεύω ότι το θέμα της ενέργειας, της παροχής ενέργειας είναι εθνική αρμοδιότητα, όχι η αρμοδιότητα της ΕΤΕ. Και όταν η ΕΤΕ επενδύει σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν άνθρακα, είναι μια στρατηγική ε, η οποία δεν είναι σωστή και δεν είναι και περιβαλλοντικά υπεύθυνη. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν εάν τα επόμενα δέκα χρόνια θα καταφέρουμε να κάνουμε μια συνετή ενεργειακή αλλαγή, όπως λέμε. Και ποιος είναι ο ρόλος που μπορούν να παίξουν οι εναλλακτικέ πηγές ενέργειας και το φυσικό αέριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα διαβάσω τον κατάλογο για να ξέρετε ποιος θα μιλήσει. Θεόδωρος. Στόλογιαν, ευχαριστώ. Μία σύντομη και τεχνική φύση ερώτηση. Από τη στιγμή που η ΕΤΕ δεν είναι κερδοσκοπική τράπεζα όπως προβλέπει το καταστατικό, ε, προς τι αυτή η ισόρευση κερδών όπως είπατε και ε, συσσόρευση κερδών που μάλιστα τα κράτησε η τράπεζα, δεν τα μοίρασε στους μετόχους. <laughs> Όντως ήταν πολύ σύντομη και αφήσει η ερώτηση. Η Σιλβή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χόριερ. Γεια σας, καλημέρα σας, χαίρομαι που είμαι εδώ. Θα ρωτήσω στα γαλλικά. Λοιπόν, αν οι πληροφορίες μου είναι σωστέ το 2005-2006 η ΕΤΕ είχε βγάλει μετοχές ε, στην αγορά εσείς ε, για να κερδίσει χρήματα. Εσείς ε, φανταστήκατε να κάνετε κάτι τέτοιο σε μία φάση όπου ε, δεν έχουμε πολλά κεφάλαια που κυκλοφορούν ε, και σε αυτή τη φάση επίσης όπου η αποταμίευση είναι αρκετά ψηλή στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Τσάρον, τρεις σύντομε ερωτήσεις. Καταρχάς αναφέρατε την καλή κατάσταση της ΕΤΕ. Αυτό σε τι οφείλεται, στην, ε, στην απόδοση, στα κρατη μπορείτε να αποδώσετε την ε, τράπεζα, μάλλον να την, ε, να την ε, χρησιμοποιήσετε ως σημείο αναφοράς για τα ευρωομόλογα, διότι συζητούμε πολύ συχνά στο Ευρωκοινοβούλιο για τα ευρωομόλογα και για τη διαφορά των spread στην Ευρωζώνη. Και πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να εξομαλυνθεί αυτή η διαφορά των spread. Έπειτα, στα projects, στα έργα, πώς ε, διενεργείτε ελέγχους, πότε είστε ευχαριστημένοι με ένα project, έχετε μακροοικονομική ε, αξιολόγηση. Τι γίνεται λοιπόν με τους ελέγχους και ποιο ποσοστό των έργων σας, των έργων που χρηματοδοτείτε είναι επιτυχές. Τρίτη ερώτηση. Ποια είναι η θέση της ΕΤΕ στην ε, EBRB με το Λονδίνο θεωρείστε ανταγωνιστές, ε, συμπληρώνει το ένα όργανο το άλλο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ε, ευχαριστώ πολύ. Βίκη και μετά βλέπω ότι και ο κύριος Όντι θέλει κάτι να σχολιάσει. Βίκη, ευχαριστώ πολύ κύριε Χόριερ. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας είπατε πόσο σημαντικό είναι να αρνείστε τη χρηματοδότηση σε κάποια project όταν αυτά δεν είναι ε, κατάλληλα και σε αυτό οφείλεται και η καλή σας φήμη έτσι και αλλιώς. Όσον αφορά τις τετροπολογίες, οι τράπεζες που συγχρηματοδοτήθηκαν από εσάς θα είχαν ε, μικρότερη ε, αξιολόγηση κινδύνου. Και ελπίζω να το υποστηρίξετε. Δεν το έχουμε συζητήσει ακόμα στον τριμερή διάλογο, αλλά είμαι σίγουρη πως αυτό θα έρθει. Αν συμφωνήσουμε για το CRD. Όσον αφορά το ομόλογα έργου, ε, είχα πολύ θετική αντιμετώπιση, αλλά θα ήθελα να διασφαλίσω ότι ισχύει αυτό για όλα τα κράτη-μέλη. Για τη χώρα μου, τα έργα αυτά είναι πάρα πολύ ωφέλιμα για την αγορά και κάθε φορά που ρωτώ πίσω στη χώρα μου γιατί κάνετε αίτηση στην ΕΤΕ για χρηματοδότηση μου απαντούν ότι πολλές φορές δεν είναι τόσο εύκολο γιατί η τόκοι είναι υψηλή. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ε, ζητήσω και, από εσάς και από τους ε, συνεργάτες σας να συνεργαστούμε. Γιατί τουλάχιστον στη δική μου χώρα ε, θεωρείται, υπάρχει εντύπωση ότι η ΕΤΕ δεν είναι το καταλληλότερο όργανο για το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν υπάρχει καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ, Jean-Pierre Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και συγγνώμη που καθυστέρησα. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε για την προσοχή σας προς το Κοινοβούλιο διότι τίποτα δεν σας υποχρεώνει να έρχεστε. Εσείς προεδρεύετε ενό οργανού που είναι περισσότερο διαθεσμικό και όχι θεσμικό. Εμείς, ένα εμείς ε, έχουμε εναλλακτικά ένα χρόνο, ναι ένα χρόνο όχι, στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού κάνουμε την έκθεση του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, εσείς δεν έχετε τραπεζική εποπτεία και ούτε έχετε ρυθμιστικό έλεγχο. Ε, εμείς ζητούμε να έχετε έλεγχο. Τι λέτε εσείς γι' αυτό, ο προκάτοχός σας ήταν υπέρ δεν πετύχαμε όμως ποτέ τον πολιτικό συμβασμό για αυτήν την εποπτεία. Τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν ιδιαίτερα την, ετο, την ΕΤΕ και φοβούμαστε μήπως χάσετε το τριπλό α. Το Κοινοβούλιο ψήφισε πολλές φορές ε, την επιθυμία του, η Ευρωπαϊκή Ένωση διορθώνομαι, θέλει να γίνει μέτοχος της ΕΤΕ παράλληλα με τα κράτη-μέλη. Τι λέτε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Οπότε δεν ξέρω αν ο εισηγητής μας ο Μάριο Μάουρο θέλει να δευτερολογήσει, να αφήσουμε όλο το χρόνο που μας έχει απομείνει στον κύριο Χόγερ για να απαντήσει. Πρόεδρε, προτιμώ να ακούσω τον πρόεδρο Χόγερ και να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές οι οποίοι είναι διαθέσιμοι να συνεργαστούν για το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει στις 10.30 να περάσουμε στη συζήτηση του επόμενου θέματος. Έχει απομείνει ένα 20 λεπτό, οπότε έχετε το χρόνο να αναπτύξετε και πιο διεξοδικά θέματα που έμειναν και από πριν ενδεχομένω. Δεν θα καταφέρω να απαντήσω σε όλα, μακάρι να μπορούσα. Γι' αυτό θα προσπαθώ. Θα απαντήσω όμως γραπτά. Αυτό σας το υπόσχομαι. Για παράδειγμα για την ερώτηση της κυρία Γκουλάρ. Είναι ε, πολλές λεπτομέρειες για να απαντήσω τώρα προφορικά. Θα τις απαντήσω γραπτά. Όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική, αυτό είναι ένα ζήτημα που συζητείται γενικότερα για το μέλλον της ενεργειακής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναφέρθηκαν και οι θέσεις σας εδώ και η τράπεζα βρίσκεται σε δύσκολη θέση διότι Έχουμε 27 αφεντικά στην ουσία από κάθε κράτος μέλος και αντιπροσωπεύουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις. Βέβαια, η τράπεζα όσον αφορά την ενεργειακή και κλιματική πολιτική έχει τη δική της ατζέντα. Περίπου πριν από 10 χρόνια είχαμε λιγότερο από 100 εκατομμύρια στη διάθεσή μας για περιβαλλοντικά έργα. Τώρα είναι, έχουμε δισεκατομμύρια για τέτοια έργα στη διάθεσή μας. Έχει γίνει μια μεταφορά δηλαδή, μια μετάβαση προ πιο περιβαλλοντικά έργα. Ή, ε, όμως πρέπει μαζί με εσάς, με την ε, Κομισιόν και με το Συμβούλιο να συζητήσουμε ακριβώς για τη γραμμή που θέλουμε να τηρήσουμε και να τραβήξουμε ανάμεσα ε, όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική. Είναι μια βασική θεμελιώδης απόφαση Όσον αφορά τώρα την ερώτηση για τα εργοστάσια ε, που χρησιμοποιούν άνθρακα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι σε κράτη που έχουν εξαιρετικά... να βοηθήσουμε τα κράτη που βρίσκονται σε εξαιρετικέ ε, δυσχερείς ε, συνθήκες και προσπαθούμε να εξυγχρονίσουμε τα εργοστάσια αυτά, ακόμα και τα εργοστάσια που χρησιμοποιούν άνθρακα για παραγωγή ενέργειας. Είναι σίγουρα περίπλοκο και δύσκολο το ζήτημα. Δεν μπορώ να, αυτή τη στιγμή να, σας, ε, να πω ότι αντιπροσωπεύω μία ξεκαθαρή θέση, γιατί το θέμα ακόμα είναι, είναι ρευστό και είναι περίπλοκο. Φυσικά και η τράπεζα έχει, έχει διαθέσει αρκετά κεφάλαια. Και με ρωτήσατε τι μάθαμε, τι μαθήματα πήραμε ότι, πρέπει να εργαστούμε περισσότερο, ότι πρέπει να κάνουμε καλύτερες αξιολογήσεις, να προσέξουμε επίσης, ώστε να κάνουμε καλύτερες αναλύσεις επιρρογνωμόνων προτού προχωρήσουμε στην χρηματοδότηση ορισμένων project. Χρειαζόμαστε αυτό που λέμε vigilance, διεξοδικότητα. Ε, όσον αφορά τώρα το ερώτημα για την πρόσβαση σε ρευστότητα, ε, μπορώ να σας δώσω το νομικό κείμενο που έχω στη διάθεσή μου, το οποίο είναι... για μένα είναι σημαντικό η ΕΤΕ να έχει πρόσβαση ε, ρευστότητας προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και αυτό θα σημαίνει και μια καλή και σίγουρη θέση όσον αφορά τις αγορές. Χρειαζόμαστε Εγγύησης. σαφώς. Βέβαια αυτό η θέση δεν είναι λεξεμένη σε πέτρα, ακόμα βρισκόμαστε σε προπαρασκευαστικό στάδιο και έχουμε πολλά στα οποία θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Έχουν γίνει πάρα πολλές προτάσεις. Πριν αναλάβω την ε, θέση που έχω τώρα, το ζήτημα αυτό απασχολούσε και τον ε, προκατοχό μου. Εάν η ΕΤΕ μπορεί να έχει μία λειτουργία ως ε, δεύτερη, ως, ως έσχατη λύση, ως δεύτερη έσχατη λύση. Και εδώ θα σας πω το εξής, ότι όσο έχω αυτή την ε, αρμοδιότητα θα το αρνηθώ, διότι εάν μειχθούμε σε αυτό θα υπερεκτιμήσουμε τις δυνατότητές μας και θα μπούμε σε θα μπούμε σε καταστάσεις που δεν πρέπει να αναμειχθούμε. Και θα αλλάξει εντελώς και το προφίλ της τραπεζάς μας, το επιχειρηματικό μας μοντέλο στην ε, κεφαλαιακή αγορά. Αυτή είναι η θέση μου. Όσον αφορά την ε, αποφυγή πιέσεων. Μόνο να ελπίζω μπορώ ότι θα μας υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί έχετε ανοσία από τις εθνικές πιέσεις, όπως φαίνεται. Ελπίζω λοιπόν να μας το μεταδώσετε και εμάς αυτό. Ε, η συμφωνία με την Ελλάδα τώρα. Ναι, φυσικά. Τώρα θα μιλήσω αγγλικά. Βέβαια. Θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτή την συμφωνία. Και σας διαβεβαιώ ότι ποτέ δεν συμμετείχα σε ένα παιχνίδι αμοιβέ επίρρηψη ευθυνών μεταξύ των ελληνικών αρχών της Τρόικα, του κυρίου Ράχενμπαχ, των Εθνικών Κοινοβουλίων και της Τράπεζας. Δεν έχει νόημα αυτό το παιχνίδι που ένας ρίχνει τις ευθύνες των άλλων. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε λογικές λύσεις για τα προβλήματα, σε μια υγιή βάση. Και γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι έχει χαθεί πολύς χρόνο στην Ελλάδα και φέτος με δημοψήφισμα που τελικά ήταν άχρηστο, πρώτες εκλογές, δεύτερες εκλογές. Έχουμε μια, είμαστε πια σε μια νέα φάση και μια νέα βάση διαπραγματεύσεων με, τις, με τις ελληνικές αρχές. Αυτή, αυτή τη στιγμή σας διαβεβαιώ ήταν πολύ επιτυχημένες μέχρι τώρα συνομιλίες και θα συνεχιστούν. Και Φαντάζομαι ότι θα έρθει και σε κατάθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνένεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στο πακέτο που αφορούν τον ανταγωνισμό, οπότε θα πρέπει να δώσει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα έχουμε σχεδόν άμεση εκταμείευση. Είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσουμε και αυτό που ε, είπαμε. Αλλά θέλουμε σαφή δέσμευση τη ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό ισχύει και για τα σχέδια υποδομών. Τα έργα υποδομών έχουν δύο βασικά προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι εκρεμούν μερικά σχέδια δικών δικτύων στην Ελλάδα που θα πρέπει να επαναξεταστούν από την άποψη της οικονομικής βιωσιμότητας. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, κάποιες αμφιβολίες που θα πρέπει να διασκεδαστούν. Και έχουμε και, μια περίπλοκη σχέση, ε, δομή σχέσεων μεταξύ των εργολάβων, της ελληνικής κυβέρνησης και ημών. Και για να είμαι ειλικρινής, αυτή η κατάσταση είναι πραγματικά εφιαλτική. Γι' αυτό είπαμε στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Χατζηδάκη ότι θέλουμε η ελληνική κυβέρνηση να μας βοηθήσει αν ε, θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα σχέδια. Άμεση σχέση και εγγύηση από την ελληνική κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλός ο τρόπος. Πέραν τούτου έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα, όπου εκεί μπορεί να μας βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την τελευταία διετία διαπιστώσαμε ότι είναι πολύ δύσκολος ο επαναπρογραμματισμός των διαρθρωτικών κονδυλίων. Και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε τώρα που ετοιμάζουμε τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές και το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί πραγματικά είναι ζωτική σημασία να μπορούμε να περάσουμε από θέματα που ήταν χρήσιμα πριν από μια δεκαετία σε κάτι που είναι χρήσιμο τώρα. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ήταν πολύ δύσκολο, για να μην πω αδύνατο, να περάσουμε σε έξυπνα ενεργειακά σχέδια, για ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, για ενεργειακή αποδοτικότητα στι διάφορε περιφέρειε. Γιατί ε, τα κονδύλια πηγαίνουν στι περιφέρειε από τα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά κυρίω για οδικά δίκτυα. Για θέματα μεταφορών κυρίω. Και είναι πολύ χρονοβόρη διαδικασία ε, για να βρούμε συμφωνία και να ε, περάσουμε από παλαιομοδίτικα σχέδια οδικών ε, μεταφορών σε πολύ καινοτόμα και πολύ πιο αποτελεσματικά περιβαλλοντικά και ενεργειακά έργα και σχέδια. Και ίσως εκεί στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ε, ε, Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούμε να αποκτήσουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα στον επαναπρογραμματισμό των σχεδίων. Τώρα, δυνατότητα απορρόφησης. Όντως υπάρχει πρόβλημα σε κάποιες χώρες και ο καθένας ξέρει τι γίνεται στην πατρίδα του. Θα πρέπει, πιστεύω, να δούμε εδώ τα τρία στοιχεία της ε, κοινωτικής πολιτικής από κοινού. Να τα θεωρήσουμε από κοινού. Αν θέλουμε να βελτιωθεί η δυνατότητα απορρόφησης με περισσότερο δανεισμό, θα πρέπει να έχουμε περισσότερο blending, περισσότερη ανάμειξη και περισσότερη παροχή τεχνικών συμβουλών. Αυτό θα αποτελέσει βασικό στοιχείο του έργου μας. Οπότε, τώρα που πλησιάζουμε σε, μια πολύ σε ένα πολύ φιλόδοξο προγραμματισμό για το 2012 και αύξηση των αρμοδιοτήτων ε, μας και το 2013 μετά το φιλόδοξο αυτό σχέδιο, δεν μπορούμε να μείνουμε στα ίδια. Θα πρέπει να είμαστε πιο δυναμικοί στην αγορά, πιο καινοτόμα σχέδια και έργα, εργαλεία για να μπορέσουμε στα τέλη του 2013 και μετά να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Οπότε θα πρέπει να ενισχύσουμε και την συμβουλευτική μας ικανότητα. Αυτό ήδη είναι σημαντικό στοιχείο της, του έργου μας. Δηλαδή να προσθέτουμε την παροχή συμβουλών στο lending και blending, στο δανεισμό και στην ρύθμιση και ανάμειξη. Αλλά και εκτός της τράπεζας, είπα, έχουμε σημαντικό ρόλο της ΕΤΕ. Και μάλιστα ε, είδα στις θερινές διακοπές ε, δύο ε, σχέδια πολύ μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως σχέδια περιβαλλοντικά, ενεργειακά, υποδομών. Και είναι πραγματικά σημαντική επιτυχία και της ΕΤΕ και του Περιβαλλοντικού Ταμείου, του Αναπτυξιακού Ταμείου, συγγνώμη. Τώρα, Μεσόγειος και Ανατολική Ευρώπη, δύο πολύ καλά παραδείγματα. Στη Μεσόγειο ως ε, Ευρώπη έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις, θα πρέπει να τις στηρίσουμε. Είχαμε ε, σε πολύ δύσκολες ε, συνθήκες την συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας και θα συνεχίσουμε την καλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την BERT. Ο κύριος Κλίντς έθεσε και μια ερώτηση για την BERT η ΕΤΕ είναι μέτοχος στην BERT, στην Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και οι ε, άλλοι μέτοχοι είναι και κοινοτικοί και εξοκοινοτικοί. Οπότε έχουμε μία δέσμη στόχων που δεν συνάδουν κατά ανάγκη με όλους τους στόχους της ΕΤΕ, γιατί η ΕΤΕ έχει διαφορετικούς στόχους, είναι πιο προσαρμοσμένη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε ό,τι αφορά την τήρηση των κοινοτικών διαδικασιών και των κριτηρίων, επίση υπάρχει διαφορά, γιατί στη Νέα Ζηλανδία, στην Αυστραλία, στη Ρωσία, στι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, δεν αισθάνονται οι εταίροι μα υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν και να σεβαστούν τι ίδιε αρχέ που σεβόμαστε εμεί απέναντι στο ελεκτικό συνέδριο. Εκεί υπάρχει μια δυσκολία λόγω τη διαφορά και θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη σε ό,τι αφορά τη σχέση μα και την αλληλεπίδρασή μας με την ΕΤΑ, την BERT. Πάντως, όταν ε, έπεσε το δίχως του Βερολίνου και όταν επανενώθηκε η Ευρώπη, η ΕΤΕ δεν ήταν έτοιμη τότε. Γιατί κανονικά τότε η ΕΤΕ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έπρεπε να αναλάβει την πρόκληση στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν ήταν έτοιμη όμως να αναλάβει τέτοιο έργο, λάθος κατά τη γνώμη μου. Οπότε εμφανίστηκε η ΜΠΕΡΤ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Ας μην επαναλάβουμε το ίδιο λάθος για τη Μεσόγειο. Έχουμε αγαστή συνεργασία λοιπόν με την Μπέρτ και με τον καινούριο πρόεδρο και με τον παλιό. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Τους συνάντησα στο Λονδίνο τον πρόεδρο την περασμένη εβδομάδα και προσπαθούμε να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας στην Ελλάδα ιδιαίτερα γιατί Σίγουρα αυτό που δεν χρειάζεται η Ελλάδα είναι μη συντονισμένες προσφορές και οικονομικές και τεχνικής αρρωγής. Θα πρέπει να έχουμε συντονισμό και η ιδιωτικοποίηση είναι κάτι που μπορεί να το κάνει καλύτερα η BERT. Σε ό,τι αφορά τη παροχή τεχνικών συμβουλών, καλύτεροι είμαστε εμεί, η ΕΤΕ. Από το συντονισμό θα κερδίσει η Ελλάδα, από τι κοινέ προσπάθειες. Γι' αυτό και συμμετέχουμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο τη ΕΤΑ. Γι' αυτό το έργο μα δεν μπορεί να είναι αντιφατικό ή ανταγωνιστικό. Θα πρέπει να επιδιώξουμε τη συνεργασία και το συντονισμό. Τώρα, Κύριε Λάγκεν, μεγάλη έκθεση της ΕΤΑ στο Νότο. Αυτή είναι η ισορροπία την οποία πάντα πρέπει να προσέχουμε. Ο στόχος της ε, ΕΤΕ είναι καθορισμένος βάσει συνθήκης και ο στόχος έχει να κάνει με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συνοχή. Η συνοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική και η εξισορρόπηση των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι το έργο μας. Και υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει, υπάρχουν ανισορροπίες που πρέπει να διορθώσουμε. Αυτό είναι το έργο μας εξάλλου. Από την άλλη, η ΕΤΕ είναι η τράπεζα των 27 και των 28 σύντομα. Δεν γίνεται αλλιώ. Δηλαδή, φανταστείτε, τον τελευταίο χρόνο πέρασα την ώρα μου συζητώντας με και προσπαθώντας να πείσω τους Υπουργούς Οικονομικών για την αύξηση κεφαλαίου. Δηλαδή φανταστείτε να τους έλεγα θα ήθελα πάρα πολύ 1,6 δισεκατομμύρια, αλλά δεν πρέπει να ενοχλήσω, ε, για παράδειγμα, τους ε, Βρετανούς ομολογούς μου για αύξηση κεφαλαίου. Καταλάβετε, είμαστε η τράπεζα των 27, των 28. Δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε προτιμησιακές ε, χρήσεις των κεφαλαίων, όπως... Ε, και αυτό θα, με αυτό θα απαντήσω και στην ε, συνάδελφο από τον Ινωμένο Βασίλειο που διατύπωσε την σχετική ερώτηση αυτή. Ναι, πραγματικά πρέπει να μιλήσουμε κύριε Χόιερ. Είμαι έτοιμος. Τώρα όσον αφορά τις προτεραιότητες που έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Πιστεύω πως είναι προφανές ότι η ΕΤΕ έχει τεράστια επενδυτική ε, δυνατότητα, αλλά πρέπει να, δια... να τηρήσει τις ε, κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση για τις ε, δυνατότητες αυτές. Εμείς πιστεύουμε ως ότι ο ρόλος της Ευρώπης ε, στην παγκοσμιοποίηση πρέπει να ενδυναμωθεί. Και αν αυτό γίνει σωστά και θα μπορέσουμε να δούμε και τα προβλήματα και τις ελλείψεις που έχουμε. Εάν εμείς είμαστε έτοιμοι να δράσουμε με την, μαζί με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ταυτόχρονα ξέρουμε ότι η ενεργειακή αλλαγή μπορεί να συμβεί μόνο εάν χρησιμοποιήσουμε έξυπνους πόρους. Και αυτή είναι μια επένδυση που έχει όγκο τον οποίο δεν μπορεί να επομιστεί ένα μόνο κράτος μέλος. Πρέπει να το κάνουμε αυτό συνολικά και με συγκεκριμένε προτάσεις. Και θα το κάνουμε. Και φυσικά κάποια από αυτά τα ζητήματα δεν έχουν άμεση προτεραιότητα διότι τα εν λόγω κράτη-μέλη δεν έχουν καταφέρει να εντάξουν στο δικό τους εθνικό νομικό πλαίσιο την ενεργειακή αλλαγή έτσι ώστε αυτή να μπορεί να πραγματοποιηθεί. Και τέλος επιμένω, η οικονομία του χώρου της γνώσης. Κάνω πολλές ε, παρουσιάσεις για αυτό το θέμα και επιμένω για την αναγκαιότητα των επενδύσεων στην καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη. Αν δείτε, η κατάσταση είναι τραγική ανάμεσα στα κράτη-μέλη στον ε, τομέα αυτό και εμείς ελπίζουμε να μπορέσουμε να προσφέρουμε βοήθεια για να αντιμετωπίσουμε την ε, πρόκληση της παγκοσμιοποίησης. Επίσης, ο έλεγχος είναι κάτι αρκετά δύσκολο. Πρέπει να το ζυγίσουμε, να το ζυγιάσουμε αυτό ανάλογα με προς τις υποχρεώσεις μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να δείτε ότι τα project ανά την Ευρώπη είναι πολλά και διάφορα. Κάποια έχουν αρχίσει 15 χρόνια πριν. Μπορείτε να, να αναρωτηθείτε για κάποια από αυτά, μα πώς είναι δυνατόν να εγκρίναμε κάτι τέτοιο. Αλλά καταστάσεις, οι συνθήκες αλλάζουν και αν γίνει ένα λάθος πρέπει να μάθουμε από αυτό και να μην το επαναλάβουμε. Και έπειτα, εάν συμβεί κάποιο λάθος, τότε οι τράπεζες οφείλουν να προασπίσουν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα... Και στην περίπτωση ενός έργου που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, πρέπει να μπορούμε να πούμε ότι η τράπεζα δεν έχει επιβαρύνει τους φορολογούμενους, δεν έχει καταγράψει ε, ζημίες, δεν έχουν πάει όλα τα χρήματα χαμένα. Φυσικά δεν είμαστε μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ε, είμαστε μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αλλά πρέπει να προσέξουμε, να ελέγξουμε και να διαχειριζόμαστε καλά το αποθεματικό μας, το οποίο έχει αυξηθεί, είναι πέντε φορές μεγαλύτερο από το κεφαλαίο που επένδυσαν τα κράτη-μέλη αρχικά. Προσπαθούμε να κάνουμε μεγιστοποίηση του κέρδου. Τώρα, από ό,τι μου λένε, πρέπει να προχωρήσω. Αλλά κάτι τελευταίο και πάρα πολύ σύντομο όσον αφορά την αποπτία. Και την συζήτηση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα στο ΕΚΟΦΗΝ για την Τραπεζική Ένωση και τα όργανα που χρειαζόμαστε. Εμείς είμαστε απόλυτα ανοιχτοί. Είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι με το ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας στο Λουξεμβούργο και συνεργαζόμαστε άριστα με τους Ευρωπαίους συντονιστές, αλλά εάν η ΕΚΤ θέλει να τραβήξει όλες τις αρμοδιότητες προς τα κίνη, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε μορφή συνεργασίας. Τα υπόλοιπα σας υπόσχομαι, θα σας τα απαντήσω γραπτός. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς, Βέρνερ, πρέπει να συνεχίσουμε στο επόμενο θέμα. Εκτός αν είσαι πάρα πολύ σύντομος πραγματικά. Γραπτή ερώτηση. Η ΕΤΕ έχει μια τεράστια δυνατότητα για να αξιολογήσει, την οικονομική, να αξιολογήσει οικονομικά τα διάφορα project. Εκτός από αυτά υπάρχει, ε, υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής ε, εταιρείας αξιολόγησης. Όχι, απαντά ο κύριος Χόιερ κατηγορηματικά. Μάλιστα, ήσταν σύντομος, αφέστατος. Υπάρχει, αν υπάρχει κάτι που δεν σας έχει απαντήσει ο κύριος Χόιερ και θα ήθελατε να του το θυμίσω, τότε πραγματικά ε, ε στείλτε μας ένα σημείωμα γραπτός. Right, we are going to move straight. Προχωράμε ακάθεκτη στο επόμενο σημείο της ημερήσης διάταξης, το 16, που όπως ε, σας είπα θα συζητηθεί πριν το 15, πριν την έκθεση Tyson. Παρακαλώ όσοι βγαίνουν από την αίθουσα να το κάνουν σιωπηλά. Τη συζητήσει εκτός αίθους παρακαλώ. Περνάμε λοιπόν στι ποινικέ κυρώσει για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικέ πληροφορίε και τις πράξεις χειραγώγηση αγοράς Η συγκήτρια μα υποσχέθηκε ότι δεν χρειάζεται πολύ χρόνο, θα τη δώσω το λόγο και περιορισμένο χρόνο αγόρευση. Παρακαλώ, οι συνομιλίε και τα πηγαδάκια εκτό τη αιθούση. Δεν μας περισσεύει χρόνος. Um, Ευχαριστώ. Είπα ότι δεν χρειάζομαι πολύ χρόνο. Κυρίως γιατί για τα περισσότερα αυτά θέματα οι τροπολογίε βελτίωσαν το κείμενο, ήταν πολύ καλές και εξαιρετική συνεργασία και με τους σκιώδεις ηγητές. Μία σύντομη ενημέρωση θα σας κάνω, Σάρων. Είχαμε δύο συνεδριάσεις των σχεδόν εισηγητών. Έχουμε καταρτήσει και τις συμβαστικές τροπολογίες. Οι σκιώδεις εισηγητές υπέβαλα κάποιες τεχνικές ε, τροποποίησεις ε, και κάποιες ερωτήσεις, αλλά είμαστε έτοιμοι ε, για τις ψηφοφορίες. Και ευχαριστώ τους συναδέλφους για την αγαστή συνεργασία, για τις ιδέες τους, τις τροπολογίες τους. Καλύψαμε και το θέμα των, οροσο... των των συγκριτικών κανόνων, το πρόβλημα των διατραπεζικών επιτοκίων Libor ε, και Euribor και θα συνεχθούμε και με τον Επίτροπο Μπαρνιέ για να συμφωνήσουμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό πριν να ξεκινήσουμε τους τριμερείς διαλόγους και τις διαπραγματεύσεις. Πάντως βρισκόμαστε στο ίδιο μήκο κύματο και χαίρομαι. Έχουμε προγραμματίσει και την ακρόαση και θα ήθελα να είναι αθρώα η προσέλευση. Ε, εντυπωσίασε που ο Γκάρι Γκάνστερ θέλει να συμμετέχει με βίντεο διάσκεψη θα έχουμε τους επιτρόπους Μπαρνιέ και Αλμούνια, θα είναι πραγματικά υψηλού επίπεδου αυτή η διάσκεψη, γιατί μας ενδιαφέρει να βρούμε τα benchmarks, τους συγκριτικούς κανόνες και είναι θέμα συναφές με το αντικείμενο της ακρόασης. Τελικίες συμβαστικέ προτάσεις. Βέβαια, θα, σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να ξανανοίξουμε τη διορία για τις τροπολογίες και να έχουμε συνεργασία με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Συναντήθηκα και με τον ε, εισηγητή της Γνωμοδότης. Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές και μετά από διαπραγματεύσει που έκανε η Σάρα, έχουμε κοινέ αρμοδιότητε, επιμερισμένε. Καλύτερα να καταλήξουμε συμφωνίε παρά να έχουμε ψηφοφορίε αντιφατικέ. 58 τροπολογίε, 18 από την Επιτροπή ΛΙΜΠΕ και οι δικοί μα συνάδελφοι τη δική μα Επιτροπή ε, ευθυγραμμίστηκαν με, την, ε, με τον κανονισμό για την αποφύγη κατάχρηση τη αγορά. Επίση, ε, κάποιοι ορισμοί από τον από τον κανονισμό μπήκαν στην οδηγία. Ε, είχαμε πολλές τροπολογίες για τη χειραγώγηση των benchmarks. Τη συμπεριέλαβα σε μια συμβαστική τροπολογία για να ε, διαμορφώσουμε ένα σαφές νομικό κείμενο. Ένα άλλο θέμα, ε, τροπολογία ΣΥΡΠΑ Πετικάνεν. Θελήσαμε να το καλύψουμε για κάποιον που, συστήνει ή παρατρύνει κάποιον να ξεκινήσει μια συναλλαγή, να καλύπτεται και αυτό το θέμα από την οδηγία, όπως καλύπτεται από τον κανονισμό. Αυτό που πρόσθεσαν οι συνάδελφοι της Επιτροπής ΛΙΜΠΕ είναι ότι θέλουν ε, ε, ελάχιστο και ανώτατο όριο, τουλάχιστον πέντε, χρόνια για τέτοιε ε, δυσυναλλαγέ ανθρώπων που κατέχουν πιστευτικέ πληροφορίε και δύο χρόνια για διάδοση πληροφοριών με σκοπό τη χειραγώγηση αγορά ε, από ανθρώπου που κατέχουν πιστευτικέ πληροφορίε. Καταρχήν θα μπορούσα να δεχτώ τι τροπολογίε, γιατί θέλω να είμαστε σαφεί ότι αν θέλουμε αρμονισμένο καθεστώ και αρμονισμένη προσέγγιση για να πατάξουμε τη χειραγώγηση τη αγορά και τη καταχρήση, θα πρέπει Φυσικά αποκλείται να έχουν όλα τα κράτη τις ίδιες κυρώσεις, αλλά τουλάχιστον σε εναρμονισμένο καθεστώς να έχουμε κάποια ανώτατα και κατώτατα όρια. Επίσης, υποχρέωση των κρατών μελών ε, για κατάρτιση αστυνομικών ε, ε, νομικών και δικαστικών και βελτίωση των ανακριτικών μεθόδων, ανακριτικών εργαλείων. Βέβαια, πολλοί δεν συμφωνούν. Εγώ θέλω να γίνεται κατάρτιση για τις ε, ανακριτικές μεθόδους. Δεν λέμε ποιες ε, μεθόδους εφαρμόσουν, αλλά ότι πρέπει να βελτιώσουν την κατάρτιση για τα θέματα αυτά. Επίσης θα ξεκινήσω διμερείς συμφωνίες και με τους σκιώδεις συγκητές μου για να ευθυγραμμίσουμε την οδηγία με τον κανονισμό. Να υπάρχει συνοχή, να μην υπάρχει ασυμβατότητα. Και κάποια θέματα ίσονος σημασίας που επίσης θα τα συζητήσουμε με τους σκιώδεις Ωραία, ας περάσουμε στους κοιόδης Δεν βλέπω την κυρία Πετικάναν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που την αντικαθιστά. Εν έρθει αργότερα θα της δώσω το λόγο. Από τους φιλελευθέρους ο Βολφ Κλίντς. Δεν έχω πολλά πράγματα να προσθέσω σε αυτά που είπε η Αρλίνα. συμβαδίζουν οι απόψεις μας και την υποστηρίζουμε. Δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρειες. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και με τους άλλους και οδησυσυγητές για αυτό το ντοσιέ. Ευχαριστώ. Ο Σβέν. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ την εισηγητρία για την ε, προσέγγιση της που μας βρίσκει σύμφωνος. Επίσης σημαντικό είναι να οργανώσουμε και την ακρόαση και οι συγγήτρια και οι συγγητές να είναι ανοιχτοί προς τα αποτελέσματα και τις προτάσεις που θα προκύψουν στη δημόσια ακρόαση και να βρούμε τρόπους να τα συμπεριλάβουμε στην ε, έκθεσή μας. Αλλιώς ίσως κατηγορηθούμε ότι οργανώνουμε ακροάσεις μόνο και μόνο για το Θεαθήνα και για την προβολή και τη δημοσιότητα, αν δεν τις λαμβάνουμε υπόψη. Θα ήθελα να είμαστε ανοιχτοί και διαλλακτικοί προς τα συμπεράσματα και τις ιδέες αυτής της ακρόασης. Συμφωνούμε και με την προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την προσθήκη που προτείνει. Πιστεύουμε όμως ότι ο ορισμός του NDC καλύπτεται στην νέα πρόταση. Η νέα πρόταση στηρίζεται σε αξίες ή παράγωγες αξίες, παράγωγες τιμές που, που στηρίζονται σε επιτόκια ή τιμές. Ίσως δεν αρκεί αυτός ο, ορισμός να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή των πιθανών δικτών και να ίσως να διευρύνουμε κάπως τον ορισμό. Για τις τροπολογίες μας. Καταθέσαμε κάποιες τροπολογίες κυρίως τις τροπολογίες 42 και 55 και την 56 που προτείνουν κάποια αποσαφήνιση στην οδηγία. Θα πρέπει να πούμε ότι η ανάγκη για εθνική νομοθεσία για τις κυρώσεις θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το άμεσο ε, οικονομικό αποτέλεσμα της κατάχρησης, αλλά οποιαδήποτε στρέβλωση, στρέβλωση για τρίτους στις αγορές και γενικότερα ευρύτερα οικονομικά θέματα. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες των συναδέλφων, συμφωνούμε με πολλές από τις τροπολογίες αυτές. Πιστεύουμε ότι ε, έγιναν πολλές βελτιώσεις στον ορισμό της κατάκρισης αγοράς, ώστε να περιλάβει και τον όρο συμπεριφορά. Και ότι αυτή η συμπεριφορά θα είναι κυρώσιμη, έστω και αν είναι έμεσα η αιτία αυτή η συμπεριφορά, η αιτία της κατάχρησης, έμεση αιτία της κατάχρησης. Η κυρία ε, Σούιμπερ για την αιτιολογική σκέψη 6 νέο, συμφωνούμε να έχουμε ευρύτερο ορισμό της κατάχρησης και να είναι σαφές ότι αν υπάρχει σχέση έστω και έμεση, μεταξύ της καταχρηστικής συμπεριφοράς και του χρηματοδοτικού εργαλείου να ισχύει ο ορισμός κατάχρησης. Επίσης συμφωνώ με τις τροπολογίες 3 και 4 της ΣΥΡΠΑ Πιετικάινεν. Χαίρομαι για τα κίνητρα να ποινικοποιηθεί το insider dealing, οι συναλλαγέ μεταξύ ανθρώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και επίση το 4 συμφωνούμε ότι πρέπει να προβλεφθεί προστασία για μη θεμητή ε, αποκάλυψη πληροφοριών. Και αυτός που ε, αποκάλυψε πληροφορίες όφιλε ή έπρεπε να γνωρίζει ότι οι πληροφορίες ήταν ανακριβείς ή παραπλανητικές. Επίσης, ε, τροπολογία τρεμόσα για το άρθρο 4, ότι η καταχρηστική πώληση προϊόντων σε μη επαγγελματίες ε, επενδυτές θα μπορούσε να επισύρει ποινές, αν και αυτό είναι θέμα για την οδηγία MIFID περισσότερο. Τέλος, έχουμε επιφυλάξεις για δύο τροπολογίες. Η μία είναι η τροπολογία 23 της αξιότιμης και εξουσέφεσης συναδέλφου Σιλβί Γκουλάρ, που λέει ότι υπάρχει ένα παραθυράκι για πληροφορίες που δίνονται για δημοσιογράφους. Θα πρέπει εδώ όμως να το διευκρινίσουμε. Ναι, με να προστατεύσουμε τους δημοσιογράφους, αλλά αυτός που ίσως χρησιμοποίησε το δημοσιογράφο προκειμένου να διασπείρει είτε εμπιστευτικέ είτε παραπλανητικές πληροφορίες, αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να ε, μπορεί να προσάγεται στα δικαστήρια ή ε, ε, το επιβάλλονται κυρώσει. Αλλιώ δημιουργούμε ένα παραθυράκι. Γιατί μερικέ φορέ η κατάχρηση των αγορών ε, περνά μέσα από τα μέσα μαζική ενημέρωση. Να μην αφήνουμε ένα γενικό παραθυράκι εκεί. Και για την αιτιολογική σκέψη 18, πρόταση Wolf Klintz. Διαφωνούμε με την ιδέα ότι οι διοικητικέ και ποινικέ κυρώσει θα πρέπει να αλληλοαποκλείονται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει νομικό πρόβλημα με την παράλληλη ισχύ διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. Αυτά και προσβλέπω σε συνέχιση τη αγαστής συνεργασία με την εισηγήτρια του υπόλοιπου και οδησηγητές για ένα αίσιο πέρα στις διαδικασίες. Άλλωστε υπάρχει ήδη αρκετή σύγκληση απόψεων. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιο εκ μέρου του ECR, της ομάδας ECR, κάποιο ε, για την ΚΟΕ. E? Μαρίσα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ, όπως και οι προλαλήσαντες, να ευχαριστήσω την Αρλίν για την πρότασή της και να πω ότι συμφωνώ με τις αδρές γραμμές της έκθεσής της. Και χαίρομαι που δέχτηκε πολλές τροπολογίες στην ε, έκθεσή της που ούτως ή άλλως ξεκίνησε με πολύ καλή βάση. Τελικά με τις αλλαγές που έγιναν στις επιτροπές δεν προλάβαμε να καταθέσουμε τροπολογίες, αλλά θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για το θέμα της έκθεσης. Θεωρώ ότι έχουμε τέσσερα είδη πολύ διαφορετικά τροπολογιών. Η μία φορά α, τις κυρώσεις α, κάποιων συμπεριφορών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή οδηγίες. Άλλες τροπολογίες αφορούν την διευκρίνηση των ορισμών και των διαφόρων ενιών. Μία ομάδα τροπολογιών αφορά την ε, προσθήκη κάποιων ε, συμπεριφορών που ίσως ε, θα πρέπει να υποβάλλονται σε κυρώσεις. Και έχω και κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Πιστεύω ότι αυτή η οδηγία, όπως φαίνεται και από πολλές τροπολογίες και για να είμαστε συνεπείς και συνεκτικοί με αυτό που προτείνεται, θα πρέπει να αποφύγουμε την αύξηση των εξαιρέσεων για να μην δημιουργήσουμε ένα νομοθέτημα που θα γίνει σαν ελβετικό τυρί, γεμάτο τρύπε, κάτι που θα αποβεί βάρος αποτελεσματικότητας. Γιατί μερικοί θέλουν να προσθέτουν ε, έννοιε να προσθέτουν συμπεριφορέ να αποφύγουμε τέτοια υπερβολική προσθήκη και πολλαπλασιασμό των ενιών, γιατί θα αποδυναμωθεί η θέση μας. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι θα πρέπει να τιμωρούμε προθέσεις και συμπεριφορές και όχι να τιμωρήσουμε τον ανταγωνισμό. Θέλουμε μια συνεκτική νομοθετική πρόταση που θα αποφεύγει παρερμηνίες, δεν θα περιέχει ασάφειες και θα διευκολύνει τους ε, εποπτικούς φορείς. Θα αποτελέσει δηλαδή ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εξασφάλιση ακεραιότητας της αγοράς. Αυτός είναι ο στόχος της νομοθετικής αυτής πρότασης και αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος που θα επιδιώκουν και οι τροπολογίες που θέλουν να τη βελτιώσουν. Ευχαριστώ και είμαι στη διάθεση της ηγήτριας για περαιτέρω συνεργασία. Έχω εγώ ορισμένα σχόλια. Υπάρχει κάποιο άλλος που θα ήθελε να μιλήσει πιο πριν. Μάλιστα, τότε θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με πολλές τροπολογίες. Δεν είμαι η εισηγήτρια, αυτό είναι δουλειά του Βόλφ, αλλά συμφωνώ με τον Σβέν για το ότι οι διοικητικές ποινικέ κυρώσεις δεν πρέπει να είναι εναλλακτικέ λύσεις. πρέπει να μπει κάποιο στη φυλακή. Ε, έχει νόημα. Αν κοιτάξουμε γενικά το πακέτο των ποινών, αλλά αυτό είναι κάτι ξεχωριστό και αυτό πρέπει πιστεύω να το αφήσουμε στο δικαστικό σύστημα να αποφασίσει. Ιδιαίτερα επειδή εφαρμόζονται οι κυρώσεις σε διαφορετικές περιπτώσεις, σε διαφορετικά άτομα γενικά, σε γενικές γραμμές, οι δημοσιογράφοι που αρθρογραφούν για τα χρηματοπιστωτικά, ναι, μπορούν να επηρεάσουν τις αγορές. Και οι δημοσιογράφοι πρέπει να ενεργούν προς το κοινό συμφέρον. Γι' αυτό εγώ δεν θα τους έδινα πάσο και απόλυτη ελευθερία να κάνουν πράγματα τα οποία μπορούν να βλάψουν τους επενδυτές και τις συντάξεις των ανθρώπων μόνο και μόνο επειδή δεν δέχονται την δημόσια ευθύνη που έχουν να μην διαχέουν πληροφορίες και προτιμούν αντί για το κοινό συμφέρον να κοιτάξουν την είδηση. Επίσης, συμφωνώ με τις τροπολογίες ε, που αναφέρονται ότι για τα ε, έμεσα βήματα που πρέπει να ληφθούν. και πρέπει να έχουμε ευρύ φάσμα. Χρειαζόμαστε βέβαια έναν ε, σαφή ορισμό των χρηματοπιστωτικών οργάνων, διότι εάν θέλουμε να ε, μεταφέρουμε τις αρμοδιότητες του σε κάτι άλλο, φυσικά δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Όμως πρέπει να αναλογιστούμε και τα προβλήματα τα οποία αυτό μπορεί να δημιουργήσει, αν μετατεθούν δηλαδή οι αρμοδιότητες και εάν πρέπει να καλύψουμε περισσότερα πράγματα από ότι απλά ένα benchmark, μια συγκριτική αξιολόγηση. Και πρέπει να λάβουμε και υπόψη την εμπειρία που έχουμε, που μας λέει ότι απλά ήταν τύχη αυτό που συνέβη στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ιδιαίτερα αν δείτε το αποτέλεσμα, που δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο. Αυτά είναι ολίγης από μένα. Ε, είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν επιθυμεί να λάβει το λόγο. Τότε επιστρέφουμε σε σένα, Αρλίν. Νομίζω πως ήταν πολύ χρήσιμο που είχαμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων, διότι για μένα ενισχύει απολύτως αυτό που προσπάθησα να κάνω στους ε, συμβιβασμούς δεν θα αλλάξω πάρα πολύ το κείμενο, διότι πραγματικά ε, έχουν καλυφθεί. Αλλά θα σας διαβεβαιώσω για ορισμένα πράγματα ότι θα συνεχίσουμε αυτό που ε, προσπαθήσαμε να κάνουμε, να δώσουμε έναν ευρύ ορισμό δηλαδή, για τη συγκριτική αξιολόγηση, για τους δείκτες, για τα είδη των συμβάσεων, προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε έναν πολύ ευρύτερο ορισμό του τι είναι benchmark, τι είναι συγκριτική αξιολόγηση και νομίζω πως είναι κάτι που θα χαροποιήσει τους περισσότερους από εσάς. Επίσης, όταν κοιτούσα τις 15 τροπολογίες προσπάθησα να διατυπώσω ε, τις ανθρωπολογίες με την πιο συμβιβαστική λύση που θα ευχαριστούσε τους περισσότερους, δηλαδή γιατί για, τον, ε, για τη λέξη συμπεριφορά, το behavior που αναφέρθηκε. Επίσης, η τροπολογία της K, τη λογική σκέψη 16α. Ναι, επί της ουσίας συμφωνώ, αλλά είναι Όντω κάτι πάρα πολύ περίπλοκα γραμμένο. Είναι μια σελίδα αιτιολογική σκέψη. Και φυσικά αυτό είναι επειδή εσεί έχετε απόλυτη γνώση του τομέα, αλλά δεν χρειάζεται να έχουμε μια ολόκληρη σελίδα αιτιολογική σκέψη. Να είμαστε σύντομοι. Ξέρω ότι το κάνατε αυτό για να μην υπάρξουν παρερμηνίε και συμφωνώ με το σκεπτικό, αλλά χρειάζεται να είμαστε πιο σύντομοι. όσον αφορά την οδηγία και τις καταχρηστικές ε, την Οι καταχρηστικές πωλήσει θα καλυφθούν από την οδηγία. Δεν καλύπτει όμως το, το inside trading και την ε, κατάχρηση, καταχρηστική συμπεριφορά. Θα το ταιριάξουμε λοιπόν με την οδηγία. Τώρα δύο θέματα με τα οποία, τα οποία με απασχόλησαν πάρα πολύ και θέλω να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων όσον αφορά την ε, τροπολογία για την ε, ελευθερία του τύπου. Νομίζω πως είμαστε καλυμμένοι, δεν χρειάζεται να το τραβήξουμε. Θα ήθελα να δείξω στους ε, συναδέλφους ότι το καλύπτουμε. Μπορούμε να προσθέσουμε κάποιες διατυπώσεις που θα μιλάνε για το καθεστώς το καλύπτουμε, διότι στον περασμένο κανονισμό είχαμε πάλι την ίδια συζήτηση. Μίλησα με τον ε, τότε εισηγητή, τον κύριο Γκόμπελς, με τις αντιπροσωπείες και καταλήξαμε σε μια λύση που κάλυπτε. Μίλησα και με τις νομικές υπηρεσίες, αλλά πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν θέλω να έχω όλο ένα και περισσότερες αναφορές ε, στο κείμενο για πράγματα που έχουν ήδη αναφερθεί σε έναν τομέα. Για παράδειγμα, για τα loopholes, για τις εξαιρέσεις ε, ανθρώπων. Μπορούμε να δούμε περιπτώσεις όπου όντω οι δημοσιογράφοι είχαν ανάμειξη στην ε, καθοδήγηση της αγοράς. Αλλά και πρέπει όντω να προσέξουμε για να μην τους ε, δίνουμε περιθώρια διαφυγής. Επίσης. Σε ό,τι αφορά τη σύμπτωση, την παράλληλη εφαρμογή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. Υπάρχει μια α, παρανόηση νομίζω εδώ. Η Επιτροπή Λιμπέ μας ε, είπε ότι, θέλουμε να εφαρμόσουμε ε, μια αρχή που ε, διαφέρει μεταξύ του κοινοτικού δικαίου και του αγγλοσαξονικού δικαίου. Το double jeopardy δεν σημαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι αλληλοαποκλείονται διοικητικέ και ποινικέ κυρώσει. Απλώ δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, ε, ταυτόχρονα δύο είδη ποινικών κυρώσεων. Πάντως η νομολογία του ΔΕΚ λέει ότι μπορούν, μπορούν ταυτόχρονα να επιβληθούν διοικητικές και ποινικέ κυρώσεις, αλλά όχι δύο ποινικέ κυρώσεις ταυτόχρονα. Αλλά δεν αποκλείεται η δυνατότητα επιβολής και διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. Προσοχή λοιπόν ε, να μην παρεξηγηθεί αυτή η πρόταση από την Επιτροπή Λιμπέ, γιατί μερικές χώρες το εφαρμόζουν η Γαλλία, για παράδειγμα, και άλλες χώρες έχουν ταυτόχρονα και ποινικέ και διοικητικές κυρώσεις. Δεν ε, θα πούμε εμείς πώς ε, εφαρμόζουν τα θέματα αυτά τα κρατη Σε ό,τι αφορά τη, την υπόθεση με το Λίμπορ, το διατραπεζικό επιτόκιο, κάποιες τράπεζες ήδη είχαν ε, ε, επιβάλει πρόστιμα, διοικητικές κυρώσεις, αλλά Ίσως επιβληθεί και ποινή φυλάκισης αν κάποιος διωχθεί για μια δραστηριότητα που είναι αξιόπινη με βάση το δίκαιο. Οπότε εμείς δεν θα πρέπει να αποδυναμώνουμε ε, τα νομοθετήματα για την κατάχρηση χειραγώγης αγοράς, ε, ειδικά στην παρούσα περίπτωση. Σας διαβεβαιώ ότι δεν θα υπάρχει double jeopardy, αυτό που λέμε στο αγγλοσαξονικό δίκαιο, δηλαδή επιβολή διπλών κυρώσεων. Γιατί αυτό ισχύει μόνο για τις ποινικέ κυρώσεις, για διπλέ ποινικέ κυρώσεις, όχι για σύμπτωση διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. Αυτό και ελπίζω θα έχουμε χρόνο και περαιτέρω συναντήσεις με τους σκιώδη ηγητέ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την δημόσια κρόση για το ε, διατραπεζικό ε, επιτόκιο Λίμπορ στις 24 Σεπτεμβρίου, 3 η ώρα, την επόμενη Δευτέρα δηλαδή, εγώ θα απουσιάζω, θα προεδρεύσει η Αρλίν, που είναι και η συγγήτρια της έκθεσης για τις πράξεις χειραγώγησης και κατάχρηση αγοράς. Μην ξεχνάτε λοιπόν αυτή την ακρόαση για το Λίμπορ. Και είναι πολύ ενδιαφέροντες οι προσκεκλημένοι. Φαντάζομαι θα υπάρξει ζωηρό ενδιαφέρον και από τους συναδέλφους για την παρακολούθηση αυτής της δημόσιας ακρόασης. Τώρα, το χρονοδιάγραμμα για την οδηγία. Εμείς ε, θέλουμε να ψηφίσουμε στις 8 Οκτωβρίου, οπότε να περάσει στην Ολομέλεια της 16 Ιανουαρίου. Αυτό το χρονοδιάγραμμα έχουμε για την οδηγία, που είναι κάπως διαφορετικό από το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα του κανονισμού. Α, ξέχασα συνάδελφοι προηγουμένως ότι υποβάλαμε στο ίντερνετ ε, πριν την ακρόαση ένα ερωτηματολόγιο και ήδη έχουμε λάβει ηλεκτρονικά κάποιες απαντήσεις και μάλιστα μερικές είναι πολύ λεπτομεριακές γιατί αυτό ζητήσαμε είναι διεξοδικέ. Θα σας τις στείλω, θα το ζητήσω από τη γραμματεία να σας τις στείλει πριν τη Δευτέρα για να τις έχετε εν ώψη της δημόσιας ακρόασης. Α, το έχει κάνει ήδη η γραμματεία. Και χαίρομαι που μύθηκε το παράδειγμά μας και η Επιτροπή. Και υπέβαλε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικό της ερωτηματολόγιο τα θέματα αυτά. Μια διόρθωση. Θα ψηφίσουμε μαζί και την οδηγία και τον κανονισμό στις 8 Οκτωβρίου, όχι μόνο την οδηγία. Οπότε παράλληλα ε, δρομολογούνται και τα δύο θέματα. Οπότε επαναρχόμαστε στο προηγούμενο σημείο της σημερινής διάταξης, το σημείο 15. Πρόκειται για την έκθεση Μαριάν Τάισεν, αλλά προηγουμένως έχω μία ανακοίνωση. Να περιμένω πρώτα τον Βέρνερ Λάγκερ να πει αυτό που θέλει να πει. Όχι. Η διάσκεψη Προέδρων ανέθεσε στην ΕΚΟΝ την σύνταξη έκθεσης που θα είναι η απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έκθεση του κυρίου Βαν Ρόμπαϊ για μια γνήσια ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση. Έτσι, η διάσκεψη των Προέδρων με την ανάθεση αυτής της αρμοδιότητας υπογράμμισε την ανάγκη έγκαιρης ε, ε, διαμόρφωση θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εν ώψη τη έκθεση ΡΟΠΟΗ και πριν την τελική έκθεση του Δεκεμβρίου. Το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήσαμε με την εισηγήτρια λαμβάνει υπόψη όλου αυτού του χρονικού περιορισμού και έτσι είναι πολύ ε, στενό και βραχή, γιατί λαμβάνονται υπόψη και οι ανάγκε ε, μεταφραστικέ. Ορίσαμε λοιπόν την διορία στις 24 Σεπτεμβρίου. Πολύ βραχύβια λοιπόν. Ο πρόεδρος Σούλτς έχει επίγνωση και του θέματος αυτού και του πολύ πιεσμένου χρονοδιαγράμματος και θα επιχειρήσει να διευρύνει κάπως την προθεσμία το μεταφράσεων να μην τι άλλο, ζητώντας κατεπηγόντως τη μετάφραση και η γραμματεία θα σας κρατάει μέρο για τις εξελίξεις και κατά πόσο θα ευοδοθεί το αίτημα για παράταση τη προθεσμία. Πάντως, ας θεωρήσουμε ότι η προθεσμία λήγει 24 Σεπτεμβρίου, ευελπιστώντα 5 ώρα το απόγευμα, όχι 12 το μεσημέρι, 24 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα. Ευελπιστώντα ότι θα παραταθεί εν τω μεταξύ. Και κάτι άλλο. Η έκθεση για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό που θα αναθέτει υποπτικές αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έκθεση ε, της ΕΤΑ, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, Tyson και Giggold. Επίσης θα ακολουθήσουν πολύ στενά χρονοδιαγράμματα. Η δήλωση του Ιουνίου, όπως ξέρετε, της των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης ζήτησε από την πρώτη πρώτου την ε, εφαρμογή της εποπτείας από την ΕΚΤ και δεν ήταν σαφή τα συμπεράσματα, είπε θα τα επανέλθει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πάντω τώρα έχει κυκλοφορήσει ότι από την 1η Πρώτου 2013 θα πρέπει να εφαρμοστεί. Και αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που μας δεσμεύει. Όντως ε, υπάρχει πρόκληση λόγω της στενότητας του χρόνου, αλλά θα πρέπει ε, να τηρηθούν αυτές οι προθεσμίες, ώστε αν ε, κινηθεί ε, στο Συμβούλιο, να μην μείνει πίσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν καθυστερήσει το Συμβούλιο, εντάξει. Αλλά εμείς θα πρέπει το χρονοδιάγραμμά μας να το καθορίσουμε με βάση το σενάριο το γρήγορο. Και πάλι βέβαια ε, θα έχουμε και τις περιορισμούς μεταφραστικούς. Ο Βέρνερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Όσον αφορά την διαδικασία για το χρονοδιάγραμμα, στον κανονισμό του Συμβουλίου έχουμε μόνο ε, δικαίωμα να παραβρισκόμαστε εκεί, στις ακροάσεις. Συμφωνήσαμε με τον κύριο Ντράκη να χειριστούμε όλο το πακέτο από κοινού και όσον αφορά τα ανοιχτά έργα, τις εγγύησεις για τα ομόλογα για παράδειγμα και άλλα τρέχοντα έργα, να τα χειριστούμε μαζί. Εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει και να πράξουμε, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει καμία απολύτως επιρροή στην ε, χαρέξη της πολιτικής, ενώ το Συμβούλιο, όσον αφορά, ε, κατά τη διάρκεια της ε, συνεδρίας της του στη Λευκοσία, αν κατάλαβα καλά, Είχαμε τρεις παρεμβάσεις από την Σουηδία, την Πολωνία και την Γερμανία τότε που αμφισβήτησαν πάρα πολύ το χρονοδιάγραμμα και εάν εμείς ασκήσουμε πίεση και ασκήσουμε τα, τα δημοκρατικά δικαιώματα για τα οποία αγωνιζόμαστε κιόλας θα είναι κάτι καλό αλλά δεν πρέπει να δημιουργήσουμε πιέσεις που θα επηρεάσουν αρνητικά το χρονοδιάγραμμα. Είναι πολύ δύσκολος ο φάκελος και χρειαζόμαστε το χρόνο για να τον αξιολογήσουμε σωστά. Και το Συμβούλιο έτσι κι αλλιώς, όταν εμείς βιαζόμαστε να κανονίσουμε κάτι, πάντα καθυστερεί. Γι' αυτό παρακαλώ τι προθεσμίε ιδιαίτερα για όλη την ιστορία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τι ε, γνωμοδοτήσει, να γίνει εις βάθος χρόνου, να μην βιαστούμε. Ευχαριστώ πολύ, Βέρνερ. Αυτό αφορά την έκθεση για την Τραπεζική Ένωση και όχι αυτό που συζητάμε τώρα. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν ήταν μόνο τρεις χώρες, ήταν και παραπάνω από τρεις χώρες που ζήτησαν ε, παράταση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Και ελπίζω να μπορέσουμε να πιέσουμε το Συμβούλιο για να μας πει τι θα γίνει. Προς το παρόν όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πιέζει και προσπαθεί να τηρήσει το αρχικό χρονοδιάγραμμα και φυσικά αυτό έχει πολλά, πολλές πολιτικές ε, αφορμές, αλλά δεν πρέπει να γίνει πρόδρομος για άλλες ενέργειες. Πιστεύω πως πρέπει να είμαστε γρήγοροι στη δουλειά μας, διότι όταν το Συμβούλιο... Διότι εάν το Συμβούλιο ε, καθυστερήσει, τότε μπορούμε να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε. Τα σχόλια μπορούμε να τα εξετάσουμε στη γενική συζήτηση. Πολύ σύντομα κυρία Πρόεδρε, εγώ εντάξει. Καταλαβαίνω αυτά που λέει ο Βέρνερ και χαίρομαι που για ορισμένα ντοσιέ το Κοινοβούλιο δεν δέχεται την πίεση του Συμβούλιου και για το θέμα των διορισμών ας πούμε. Αλλά το χρονοδιάγραμμα μας το επιβάλλει το Συμβούλιο ή σήμερα απλώς υπάρχει μία γεπικρατούν επικρατούν κατεπίγουσες συνθήκες στον τραπεζικό τομέα ορισμένων κρατών που δεν έχουμε καμία σχέση ούτε εμείς ούτε το, ούτε το Συμβούλιο. Δηλαδή πρέπει απλώς να δούμε κατάματα το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατάλαβα. Και είμαι και το πρώτο θύμα για το πόσο γρήγορα δηλαδή πρέπει να προχωρήσουμε. Αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό το να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με άλλα θεσμικά όργανα. Είναι πολύ σημαντικό να βγούμε από την κρίση και πρέπει να έχουμε και τις ε, ε, τα αντίστοιχα μέσα. Για όσα υπόθηκαν, αποφασίστηκαν στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μην αρκεί, αλλά είναι απαραίτητη για να έχουμε τα κονδύλια του SM και να μπορέσουμε να επανακεφαλοποιήσουμε τις τράπεζες. Δεν πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί που θα αναβάλουν. Γιατί αν μετά υπάρξουν προβλήματα χρόνου στα άλλα θεσμικά όργανα, τότε και εμείς μπορούμε να κερδίσουμε χρόνο. Εγώ είμαι υπέρ της πρότασής σας, Πρόεδρε, αλλά θα πρέπει η έκθεση να παρουσιαστεί. Σίγουρα μετά θα έχουμε τις τροπολογίες και αν έχουμε χρόνο θα παρουσιάσουμε και παραπάνω τροπολογίες. Το σημαντικό όμως είναι να έχουμε ένα ψήφισμα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συσπήρωση από γύρω. προτεραιότητα είναι να βγούμε από την κρίση και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο και με τον πιο σταθμισμένο τρόπο. Ούτως πρέπει να πράξουμε. Συμφωνώ και με σας. Μάλιστα, με έχετε μπερδέψει λίγο. Δεν ξέρω ποιο θέλει να παρέμβει, ποιο όχι. Σφέν, είσαι εισηγητή. Ήβο, σκιώδη εισηγητή, θε να μιλήσει για την Τραπεζική Ένωση. Α συνεχίσουμε λοιπόν με τη συζήτηση τη πρώτη έκθεση Τάισεν για αυτό το θέμα, Σφέν. Ευχαριστώ. Συμφωνήσαμε με τη Μαριάν για το χρονοδιάγραμμα, γιατί Πιστεύουμε ότι δεδομένης της κατάστασης το βασικό πρόβλημα είναι ότι το Συμβούλιο αφισβήτησε το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συναπόφαση, για την πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας συναπόφασης στην περίπτωση αυτή. Και για να προασπίσουμε την επίδρασή μας στο θέμα αυτό απαιτεί να διαμορφώσουμε το ταχύτερο δυνατό τη θέση μας. Το ξέρουμε και από το παρελθόν κάθε φορά που το Κοινοβούλιο πολύ πιο γρήγορα διαθετεί τις εσωτερικές του διαφορές, ενισχύει τη διαπραγματευτική του θέση απέναντι στο Συμβούλιο. Και μέχρι στιγμής έχουμε πολύ καλές επιδόσεις. Μπορεί αυτή τη φορά να έχουμε μεγαλύτερες δυσκολίες, γιατί ήδη το νιώθουμε ε, επειδή υπάρχουν μεγάλες διαφορές. αλλά πιστεύω ότι ήδη υπάρχει αρκετό επίπεδο σύγκληση μέχρι στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε, αν προχωρήσουμε ε, γρήγορα, όπω είπε η Μαριάν, δηλαδή να καταθέσουμε, να υποβάλουμε το συντομότερο δυνατό τα σχέδια έκθεση, τότε θα έχουμε και βάση για τη συζήτηση. Αν στη συνέχεια το Συμβούλιο δεν καταφέρει να είναι αρκετά γρήγορο ε, σε σχέση με αυτό που απαιτεί η κρίση, τότε συμφωνώ με τη Μαριάν ότι και εμείς θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο. Δεν θα κατηγορηθούμε εμείς ότι κολλήσει αργούμε και ότι καθυστερούμε την όλη διαδικασία γιατί εμείς φροντίσαμε με ταχύτητα να, λύσουμε, να αντιμετωπίσουμε την κρίση και να αποσυνδέσουμε το τραπεζικό χρέος από το δημόσιο χρέος, να διαρρήξουμε αυτό το δεσμό. Όσο πιο γρήγορα λοιπόν να καθορίσουμε τη θέση μας, όπως είπε και η Πρόεδρος, και όσο πιο γρήγορα κινηθούμε, τόσο το καλύτερο. Είναι σαφές βέβαια ότι και ως Ευρωπαίοι έχουμε συμφέρον να αντιμετωπιστεί η κρίση το συντομότερο δυνατόν και να διευθετηθούν οι διαφορές με τρόπο που, θα, με τρόπο που επιτάσσει η σοβαρότητα της κρίσης. Πάντως, ακριβώς για να α, υπεραμεινθούμε τις θέσεις μας και να έχουμε πραγματικά επίδραση στην όλη διαδικασία θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα γιατί η διαδικασία επιτρέπει το σεβασμό όλων των δημοκρατικών δικαιωμάτων των Ευρωβουλευτών. Υπάρχει και χρόνος για τροπολογίες, υπάρχει και χρόνος για συζήτηση. Εγώ προτιμώ να κρατήσουμε αμετάβλητο το χρονοδιάγραμμα και να ιεραρχήσουμε και τις προτεραιότητές μας σε σχέση με άλλες εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις ε, που είναι πολύ υποδέστερες σε σημασία σε σχέση με την, ε, με την έκθεση κυρίας Τάισαν ο Ήβο. Ε, eh, Ευχαριστώ. Είμαι σκιώδης εισηγητής ε, και θα ήθελα να εκφραστώ όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει πρόβλημα με αυτήν την διαμάχη μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Αλλά εμείς εξετάζουμε θέματα τα οποία έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Πρέπει να τα αναλύσουμε με ιδιαίτερη προσοχή, όπως και τις επιπτώσεις τους. Και μετά θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο εξής ότι το θέμα χρειάζεται εις βάθος συζήτηση και πρέπει να έχει δημοκρατική νομιμότητα αυτή η συζήτηση. Πρέπει να ληφθεί υπόψη και στα κράτη-μέλη, ούτως ώστε οι θέσεις αυτές να υποστηριχθούν ευρύτατα και να μην υποστούμε σοβαρές επιπτώσεις ε, σχετικά με την κοινή γνώμη. Συμφωνώ αυτό το οποίο ο κύριος Λάγκεν είπε. Λοιπόν, πιο, πιο αργά μπορεί να σημαίνει και μεγαλύτερη ασφάλεια στα αποτελέσματα. Η Ελίζα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας και να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Όντως είναι σπευσμένη η διαδικασία, είναι λίγο άρων-άρων, αλλά δεν θεωρώ ότι θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπομειστεί το βάρος καθυστέρησης, ε, να μην κατηγορηθεί ότι παρακολεί η κολλησιεργή στη διαδικασία αυτή. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες να βάλουμε τα δυνατά μας και να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα για να μην γίνουμε εμείς ε, ε, από διαπομπέως τράγος ή το πρόσχημα, η αιτία της καθυστέρησης. Τώρα, ας προχωρήσουμε στη συζήτηση. Ακούσαμε την πρόταση, Βέρνερ. Το ζήτημα είναι πώς να έχουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή εποπτεία υπό, την, προταση βερνερ το ζητημα ειναι πως να εχουμε μια ενιαια ευρωπαικη εποπτεια υπο την τον έλεγχο της ΕΚ. Πιστεύω πως το έργο μας είναι να έχουμε μια εντατική και διεξοδική συζήτηση. Αυτό θεωρώ το σωστότερο. Σε αυτόν τον κανονισμό του Συμβουλίου να κάνουμε μία ε, ακρόαση, σύντομα. Αυτό θεωρώ σωστό. Δεν είναι καμία καθυστέρηση, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει και μπορεί να γίνει έτσι κι τον Οκτώβριο. Είναι αναγκαίο, δεν είναι καθυστέρηση. Ε, εγώ δεν θέλω να έχω στη συνείδησή μου το βάρος μιας άσχημης, μιας λάθος επιλογής, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον ρόλο μας όπως πρέπει. Εάν θέλουμε να το πάρουμε το ρόλο μας στα σοβαρά, πρέπει να κάνουμε αυτό ακριβώς αυτό. Η αγροτική πολιτική εδώ και 20 χρόνια που δεν μπορούσαμε να ε, συμμετέχουμε με τη διαδικασία συναπόφασης. Είδατε τι έγινε, έχουν υπάρξει καθυστερήσεις. Γι' αυτό λοιπόν σας κάνω έκκληση να το τηρήσουμε αυτό. Ευχαριστώ. Ξέρω πως είναι κάτι που σε απασχολεί πάρα πολύ. Συμφωνώ μαζί σου πως πρέπει να βρούμε χρόνο για ακρόαση. Επίσης, να σημειώσουμε ότι τώρα ε, πιστεύω πως καλό θα ήταν να διατηρήσουμε το σύντομο χρονοδιάγραμμα για τις εκθέσεις και εκτός αν υπάρξουν κάποια νέα από το Συμβούλιο μέχρι τότε, θα γίνει η Συμβούλιο Κοφίν στις 8 Οκτωβρίου. Και πιστεύω ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει εκεί, για να δούμε τι θα γίνει με το χρονοδιάγραμμα του Συμβουλίου. Και αν εκεί υπάρχει κάποια ένδειξη ότι το Συμβούλιο θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο, τότε Μπορούμε και εμείς να το καθυστερήσουμε χωρίς να μας προσάψουν ότι φταίμε και καθυστερούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, και, το, και το Συμβούλιο λένε ότι εμείς καθυστερούμε όσον αφορά τα CRD ε, και ότι προχωρούμε σε τριμερείς διαλόγους χωρίς εντολή. Και τα μέσα για τα μέσα ενημέρωση, αυτό είναι κάτι έτσι πολύ συναρπαστικό και το χρησιμοποιούν τι καθυστερήσει μα για την οδηγία για τι κεφαλιακές απαιτήσει. Ρίχνουν σε εμά το φταίξιμο και θα ρίξουν σε εμά το φταίξιμο για πολλά λάθη που κάνουν εκείνοι. Γι' αυτό λοιπόν ας τα κάνουμε σωστά. Α αρχίσουμε γρήγορα, α είμαστε λογικοί και σόφρονε και μετά δούμε, βλέπουμε τι γίνεται. Μαριάν λοιπόν, νομίζω πω μπορώ να σου δώσω το λόγο, επιτέλου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτή την πρώτη έκθεση την μόλις αναφέρατε, τη βάλατε πολύ σωστά μέσα στο πλαίσιο της. Η διάσκεψη των Πρόεδρων μας ζήτησε να νομοθετήσουμε σχετικά. Η ΑΦΚΟ ζητάει ενισχυμένη συνεργασία. Πρέπει να πω στους συναδέλφους ότι η εντολή μας βασίζεται στο άρθρο 225 της συνθήκης, δηλαδή αυτή η έκθεση πρέπει να καταστεί νομοθετικό ψήφισμα. Στα συμπεράσματα θα πρέπει να έχουμε έναν κατάλογο προς την Κομισιόν με συγκεκριμένα ε, ε, ζητούμενα για να παρέμβει στο νομοθετικό επίπεδο. Αυτό μέσα στα πλαίσια των συνθήκων και αν κρατηθούμε στις συνθήκες. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να πούμε ότι χρειάζονται θεσμικές, ε, συνταγματικές μεταρρυθμίσεις αλλά εκεί δεν μπορούμε να ζητήσουμε από την Κομισιόν να υποβάλει προτάσεις γιατί οι διαδικασίες είναι διαφορετικές. Μας δόθηκε η εντολή πριν από το καλοκαίρι. Οι συνάδελφοι έλαβαν ένα έγγραφο εργασίας στις 3 Σεπτεμβρίου το οποίο το χρησιμοποίησαμε για τις ακουράσεις Ντράγκη Μπαρνιέ και Ρεν και βάσει των όσων ψηφίστηκαν είχαμε και τα ψηφίσματα και τις παρατηρήσεις κατά την ακρόαση. Στις 7 Σεπτεμβρίου παρουσιάσαμε ένα σχέδιο έκθεσης και εδώ πάλι χρειάστηκε να τρέξω. Πρέπει να πω ότι όλα αυτά γίνανε πάρα πολύ γρήγορα. Είχαμε τις διακοπές, χρειάστηκε λοιπόν να αντιδράσουμε γρήγορα, αλλά σήμερα έχουμε ένα έγγραφο το οποίο μπορεί να αποτελέσει βάση για τους διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου που θα πάνε στους, ε, οι τέσσερις πρόεδροι δηλαδή που θα ετοιμάσουν τη στρατηγική για την ενίσχυση μιας πραγματικής οικονομικής νομισματικής ένωσης. Έχουμε αυτό το κείμενο, εμείς είπαμε να δράξουμε αυτή την ευκαιρία και να εργαστούμε σύντομα. Η πρόταση λοιπόν είναι μπροστά σας Και σε αυτή τη βάση θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Εγώ λοιπόν προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομη. Ξέρετε την, ε, τις, συνήθειές μου. Εδώ όμως πρόκειται για κάτι το μακροπρόθεσμο. Ξέρετε το πώς ε, ε, έχει η πορεία. Πρέπει να υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις στον κύριο ε, Βαν Ρομπόη και πρέπει να είναι επίση και αυτή ενήμερη για τις ε, δικές μας θέσεις. Αναφέρω λοιπόν στα διάφορα σημεία το την επιχειρηματολογία μας και από εδώ μπορούμε να βγάλουμε ορισμένα ερωτήματα τα οποία τα ε, θα απευθύνουμε προς την Κομισιόν και να προετοιμάσουμε και την στις παρατηρήσεις μας για την έκθεση Van Rompuy που θα παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο. Να σας τα παρουσιάσω τα πράγματα λογικά. Σε μία πρώτη φάση εγώ έχω κάνει μία ανάλυση της κατάστασης και στο κείμενο λέμε ότι ζούμε στην κοινωνία της πληροφόρησης, ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ολοκλήρωση ε, έναντι των όσων συμβαίνουν σήμερα, Όλα είναι πολύ σημαντικά να έχουμε δηλαδή να πούμε κάτι στον κόσμο για το μέλλον και μακροπρόθεσμα όλο αυτό το πέρασμα να είναι καλό για όλους. Να μην είμαστε απολώς θύματα της παγκοσμιοποίησης. Είναι πολύ σημαντικό να ενσωματωνόμαστε και να ενωνόμαστε ως το δυνατόν περισσότερο. Αυτό κατέστη όμως ακόμη πιο εμφανές με την κρίση. Είδαμε πόσο ευπαθής είναι η Ευρωζώνη μέσα από την κρίση εμείς καταλάβαμε ότι η Ευρωζώνη δεν έχει όλα τα απαραίτητα μέσα για να λύσει τα προβλήματα τα οποία έχουν προχύψει κατόπιν της κρίσεως. Θα πρέπει επίσης να βρούμε εναλλακτικέ λύσεις, διότι δεν είναι πάντα δυνατόν να τα τακτοποιούμε όλα σε διακυβερνητικό επίπεδο. Είδαμε ότι έχουμε ένα σωρό αναποτελεσματικότητες και πρέπει να κάνουμε κάτι. Χρειάζεται ένας μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών με τους στόχους. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε και τη δομή αλλά και για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη η οποία έχει χαθεί διότι κανένας δεν έχει εμπιστοσύνη πλέον ούτε στην πολιτική, ούτε στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Απ' την άλλη μεριά όμως μας ζητάνε από εμά να βρούμε τις λύσεις και αυτή είναι και η δουλειά μας εξάλλου. Είναι πάρα πολύ σημαντικός επίσης ο ρόλος των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, διότι και αυτοί θα πρέπει να συνεχίσουν να υπερασπίζονται το ευρώ και πρέπει να το θυμίζουνε κάθε φορά που επικοινωνούν με τους πολίτες πρέπει κάθε φορά που υπάρχει μία διάσκεψη, κάθε φορά που έχουμε μία συνάντηση υψηλού επίπεδου, πρέπει να λένε στους πολίτες ότι θυμούνται, ε, ότι έχουν κατά νου πόσο σημαντική είναι η Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να έχουμε διαφορετικές αποφάσεις από τα όσα, ε, συγγνώμη, από αυτά που αποφασίζονται θα πρέπει να εξηγήσουν ότι εξαρτώμεθα ημένα από τους ΔΕ και τα ψηφίσματα δεν μπορούν να είναι προσωπικού χαρακτήρα. Με την κρίση επίσης διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μία διαφορά μεταξύ των περιφερειακών κρατών με, τις, με τα κεντρικά κράτη στην Ευρώπη. Χρειάζεται αλληλεγγύη και ευθύνη, αλλά θα πρέπει να είναι υπεύθυνη μεν και αλληλεγγύη δε. Τα κράτη-μέλη επίσης θα πρέπει να σεβαστούν τις δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβαν. Θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω. Πρόκειται για μια διαδικασία χρονοβόρα, αλλά θα πρέπει να υποδείξουμε ποιος είναι ο σωστός δρόμος και άμα συμφωνήσουμε στην έκθεση των τεσσάρων προέδρων, τότε θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα πάντα βήμα προς βήμα. Το πιο σημαντικό όμως είναι να βγούμε από την κρίση. Υπάρχουν διάφορες παράγραφοι για τις ε, εκθέσεις του Βαν Ρομπόη και τις αποφάσεις της διάσκεψης κορυφής. Εμείς πρέπει να είμαστε ευτυχείς που σήμερα για πρώτη φορά δίνουμε μια εντολή για ε, μακροχρόνια εργασία. Πρέπει να έχουμε διαρθρωτικά μέτρα ως στόχο. Μέτρα μακροπρόθεσμης διάρκειας αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα βράχη πρόθεσμα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Και εδώ είναι και οι αλλαγές που θα πρέπει να επιφέρουμε στην ε, συνθήκη. Πρέπει να υποβάλουμε προτάσεις σχετικά, αλλά αυτό μακροπρόθεσμα. Όταν θα έχουμε αποδείξει στους πολίτες ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να βγούμε από την κρίση και τότε μπορούμε να προτείνουμε ακόμη και τροπολογίες. Μέσα σε αυτήν την Επιτροπή συμφωνούμε γύρω από ορισμένα στοιχεία. Ολοκλήρωση, νομισματική ολοκλήρωση της Ευρωζώνης για τους 17 ίσως να χρειαστούν ειδικά μέτρα. Αλλά θα πρέπει πάντα να έχουμε τη δυνατότητα να ε, δεχόμαστε βοήθεια και από τους άλλους, δηλαδή οι 17 είναι το μήνυμο, αλλά και άλλοι πρέπει κάτι να κάνουν. Πρέπει να λειτουργεί και η εσωτερική αγορά. Όσον αφορά τώρα στην, στην Τραπεζική Ένωση, εδώ είχαμε πολλές νομοθετικές προτάσεις. Εχθές ε, μιλήσαμε για διάφορες από αυτές τις προτάσεις. Τον μηχανισμό παρακολούθησης, μηχανισμό εποπτείας. Όπως είπαν οι συγητές, ε, οι εγγύσεις καταθέσεων. Όλα αυτά όμως ε, δεν σημαίνουν ότι πρέπει να αγνοήσουμε την Τραπεζική Ένωση πρέπει να προχωρήσουμε προς την Τραπεζική Ένωση. Δεν θα πρέπει εμείς να αφήσουμε παράμερα ορισμένα στοιχεία. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να προχωρήσουμε εξετάζοντας ορισμένα ζητήματα και μετά με την έκθεση Βαν Ρομπόη να προχωρήσουμε στο μέλλον και να καταλήξουμε στην Τραπεζική Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό, ακόμη και αν έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, με αυτή την έκθεση να προχωρήσουμε ακόμη πιο μακριά, με στόχο την Τραπεζική Ένωση. Και εδώ έχουμε διάφορα σημεία. Θα ακούσω μετά και είναι οι απόψει σας, τι λέτε εσεί για την ανεξαρτησία τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Οικονομική Νομισματική Ένωση. Μετά πρέπει να λύσουμε και το πρόβλημα του φαύλου κύκλου μεταξύ δηλαδή τραπεζικής κρίσης και χρηματοπιστωτικής κρίσης γενικότερα θα πρέπει να έχουμε έναν οργανισμό εποπτείας για τις τράπεζες, πρέπει να έχουμε μία μονάδα επίλυσης των τραπεζικών κρίσεων. Και πράγματι το πεδίο εφαρμογής μίας πρότασης θα πρέπει να αποτελεί τον καθρέφτη και για την άλλη. Αν έχουμε εμεί τον μηχανισμό εγγύσεων ή το μηχανισμό για τις λύσεις, πρέπει να έχουμε όλα τα μέτρα, ούτως ώστε να μην έχουμε εντάσεις. Αν κάνουμε κάτι με την κεντρική τράπεζα θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις πάνω στην Ευρωζώνη αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη πάντα στο νου μας την ενιαία αγορά και την ελεύθερη κυκλοφορία. Εγώ ήμουν υπέρ των προτάσεων για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εγώ ήμουν υπέρ του να τις αναθέσουμε και άλλες αρμοδιότητες πλην του SM. Αλλά ξέρετε ότι υπάρχει ένταση όσον αφορά στην ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας από τη μια και από την άλλη μεριά την accountability, δηλαδή το λογιστικό μέρος και το θέμα της εποπτείας. Εμείς μπορούμε να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας για να το καταθέσουμε στον κύριο Βαν Ρομπόι. Τώρα, για τις ακροάσεις, για τους διορισμούς, για τις παρουσιάσεις απολογισμών, θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία αυτού του επιχειρήματος. Για το εφαρμοστικό πεδίο έχουμε ε, ε, την, κεντρική τράπεζα και μετά πρέπει να έχουμε 17. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να προχωρήσουμε έχοντας έχοντάς τους όλους ισότιμους. Θα πρέπει όταν δημιουργηθεί το σύστημα εποπτείας να εισάγουμε και τις άλλες χώρες. Για το θέμα <coughs> της κατάθεσης των εγγυήσεων, της προστασίας, συγγνώμη, της εγγύησης καταθέσεων, πρέπει να προστατεύσουμε τους καταθέτες ε, αλλά και τις τράπεζες τις ίδιες διότι αν μία τράπεζα βρίσκεται σε κίνδυνο τότε υποσκάφτει όλο το σύστημα και εδώ έχουμε και τους κινδύνους, τους ηθικούς κινδύνους που, τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίσουμε και οι προδιαγραφές πρέπει να είναι πολύ ψηλέ. Και εδώ έχουμε ένα σωρό προτάσεις που εξετάζονται και συζητιώνται και πρέπει να, γίνουν, να καταστούν, να μεταφραστούν όλα αυτά σε καλές νομοθετικές πράξεις θα πρέπει στο τέλος να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα εγγύησης καταθέσεων, ένα ενιαίο ταμείο. Εγώ νομίζω ότι η έκθεση Φερέιρα ζητούσε ένα χωριστό ταμείο για την εγγύηση των καταθέσεων και για τις επιλύσεις κρίσεων. Θα πρέπει να έχουμε πλειοψηφία, μετά όμως έχουμε και άλλες δυνατότητες, ring fencing και άλλες καταστάσεις. Αλλά είναι σημαντικό να έχουμε εμείς ένα ταμείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά. Προσπάθησα να συνδέσω αυτά τα δύο στοιχεία. Και για τον ενιαίο προπολογισμό. Ήδη έχουν γίνει πολλά πράγματα και γίνονται. Εμείς ε, πρέπει όμως να επιμένουμε σε αυτό το οποίο ακόμη είναι απαραίτητο. Προς στιγμή έχουμε έναν τρίλογο και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να καταλήξουμε και εμεί με προτάσεις και ο Επίτροπος ο υπεύθυνο για το ευρώ θα πρέπει να δει αν με το SME χρειάζεται και κάτι άλλο πιο δυνατό για τις, που να γιάται τη σταθερότητα της Ευρωζώνης έτσι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με την κοινοτική μέθοδο μέσα στους προϋπολογισμούς. Μετά έχουμε ορισμένες παραγράφους σχετικά με τους εθνικούς προϋπολογισμούς και πρέπει να συντονιστούμε για αυτά. Και όσον αφορά στο χρέος, το χρέος όλης της Ευρώπης και εδώ έχουμε μερικές παραγράφους και δεν θα πρέπει να βιαστούμε στις εργασίες μας γιατί διατρέχουμε κίνδυνο. Μετά έχουμε την Οικονομική Ένωση και έχουμε εδώ διάφορα διαρθρωτικά σημεία τα οποία θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε. Λέμε ότι όλοι είμαστε τμήμα της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης. Κανένας δεν πρέπει να μείνει απ' έξω. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν στα πλαίσια της οικονομίας αγοράς. Πρέπει να προωθήσουμε την ανάπτυξη και τη σταθερότητα. Μετά μιλάμε για τους φόρους. Αυτό μπορεί να ενδιαφέρει τους συναδέλφους και να τα διαβάσετε προσεκτικά. Πρέπει να έχουμε μία λογική και αιτιολογημένη φορολογική πολιτική μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε επίσης για το γεγονός ότι η κρίση μας οδήγησε σε, συζητη... σε σχετικά με την κόβερνα στη διαχείριση, αλλά από την άλλη μεριά ενίσχυσε και το αίτημά μας για δημοκρατία. Η Επιτροπή Θεσμικών Υποθέσεων θα μου δώσει δίκιο. Αλλά και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα έπρεπε να συμμετέχει σε αυτές τις συνεδριάσεις. Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή βάση με συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλες αυτές τις αποφάσεις. Διότι πρέπει να έχουμε την δημοκρατική ευθύνη για το Κοινοβούλιο και για την Τρόικα. θα πρέπει να ακούσουμε και τους εκπροσώπους της Κομισιόν για να έχουμε μία μεγαλύτερη διαφάνεια και να ξέρουμε τι γίνεται και στο ΕΚΟΦΗΝ. Εγώ έκανα ερωτήσεις, διατύπωσα ερωτήσεις προς την Κομισιόν και στα παρατήματα σχετικά με τη μελλοντική ε, νομοθετική δραστηριότητα. Περιμένω τα σχόλιά σας και ελπίζω να μπορέσω να προχωρήσουμε γρήγορα. Σας ευχαριστώ. Έχουμε πολλά δραστήρια μέλη εδώ στην Επιτροπή ΕΚΟΝ, πέραν των σκιωδών εισηγητών και ακούω συνέχεια παράπονα ότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο για τη συζήτηση και ότι το μεγαλύτερο τμήμα του χρόνου αγόρευσης ε, το μονοπολούν οι σκιώδεις εισηγητές. Θα ακούσουμε φυσικά τους σκιώδεις εισηγητές μετά τον κύριο Κουαλτιέρη που είναι ο αρμόδιος ηγητής από την ε, Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Πέντε λεπτά στον καθένα θα δώσω και για τους υπόλοιπους ομιλητές τρία λεπτά στον καθένα. Αν χρειαστεί θα εξαντλήσουμε το χρόνο με τις παρατηρήσεις ε, των μελών, αντί να ξαναδώσουμε χρόνο για να δευτερολογήσει η Νομίζω ότι προτιμάει, το προτιμάει και η συγγετρία να ακούσει τι απόψει των συναδέλφων. Πέντε λεπτά οι σκιώδει συγγετές, τρία λεπτά οι υπόλοιποι. Θα σα διαβάσω τον κατάλογο. Ο Βέρνερ Λάγκ είναι ο πρώτος, όλο τυχαίος. Έχει μιλήσει ήδη πολύ. Μετά τους ε, uh, αυτοί και όσοι προσθεθούν, αυτοί όμως μετά τους σκιώδους ηγητές. Ματάιας uh, I'm not sure whether there's anybody here from the EFD or not, and then Roberto Galtieri. So, right, Liam. Bon, je... Trois minutes. Bon, je voudrais... Τρία λεπτά. Έχω πέντε, τόσο το καλύτερο. Να συγχαρώ τη Μαριάν για το σχέδιο έκθεσης που το προετοίμασε με ιδιαίτερα σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Αλλά απαραίτητο όμως λόγω της, ε, του κατεπήγοντος της κρίσης και δεδομένου ότι θα έχουμε μία διάσκεψη κορυφής τον Οκτώβριο γύρω από την οποία δεν μπορεί να σιωπήσει το Κοινοβούλιο. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Θα προχωρήσω πολύ γρήγορα για τα ουσιαστικά σημεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τον πρώτο στόχο αυτής της έκθεσης, δηλαδή να αντιδράσουμε στην πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Του Συμβουλίου, συγγνώμη. Πρόκειται Εδώ για τη δημιουργία του Ταμείου Λύσεων του, και του Ταμείου Διαχείρισης. Το άκουσα αυτό από τη συνάδελφο Μάριαν και θα το συζητήσουμε. Δεν έχω αντιρρήσεις. Θα υπάρξει επίσης συζήτηση και για την ε, εποπτεία. Αυτή η εποπτεία όμως θα καλύπτει μόνο τη ζώνη ευρώ ή όλη την ένωση. Και αυτό θα το συζητήσουμε τώρα για την ε, Δημοσιονομική Ένωση. Ο βασικός στόχος είναι να υλοποιήσουμε αυτό το ομοσπονδιακό άλμα παράλληλα με ένα δημοκρατικό άλμα. Διότι αυτό το ομοσπονδιακό άλμα θα το κατανοήσουν άμα δεν υπάρχει το αντίστοιχο δημοκρατικό οι πολίτες ως ένα γραφειοκρατικό άλμα. Για το θέμα της συναπόφασης τώρα. Θα πρέπει συνολικά στη φάση της έκθεσης ΑΖΕΕΣ να συμμετέχουμε στην όλη, στον όλο σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τώρα ποιος είναι αυτός ο συντονισμός εκ των προτέρων εξάντε. Εξάντε σημαίνει τι. Σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να προδικάσουμε την μακροοικονομική κατάσταση της επόμενης χρονιάς μέσα σε μια κυκλική δυναμική. Σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας λοιπόν την δυναμική των επενδύσεων. Τώρα εμείς έχουμε τους χρυσούς κανόνες. Το χρυσό κανόνα, ξέρετε ποια είναι η θέση μας στη σοσιαλιστική ομάδα. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει στον υπολογισμό του ελίματος να παίρνουμε υπόψη το, τις δημόσιες επενδύσεις. Αλλά όμως στον εξάντε λογαριασμό θα πρέπει να τα παίρνουμε όλα αυτά υπόψη μας προκαταβολικά. Δηλαδή η Πορτογαλία ας πούμε μέσω του συντονισμού εξάντε επιτρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι δύσκολες καταστάσεις για τις ενδιαφερόμενες Υπάρχει και κάτι άλλο. Ο κύριος που μιλάει για έναν Υπουργό Οικονομικών που θα διαχειρίζεται έναν κεντρικό προϋπολογισμό. Μα εδώ μας τίνει πραγματικά έναν κίστρι, πρέπει να το πιάσουμε. Διότι δεν μπορούμε εμείς να μιλάμε για όλα τα προηγούμενα και να μην έχουμε από την άλλη μεριά έναν στεναρό προϋπολογισμό ο οποίος θα αναλαμβάνει πρωτοβουλία στον τομέα των επενδύσεων πράγμα το οποίο κάνανε πρώτα μονομένα τα κράτη-μέλη. Μιλήσατε για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και φορολογικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν. Αλλά πρέπει όμως να βγάλουμε και το δίδαγμα, διότι εφαρμόστηκαν μείωση της, ε, του μισθού, μείωση της ευελιξίας, ε, μείωση της προοδευτικότητας των συστημάτων συλλογής των φόρων λειτουργήσαν όλα αυτά. Αυτά είναι αμφίβολα. Το αποτέλεσμα είναι αμφίβολο. Εμείς θέλουμε μία οικονομική πολιτική όπου από τη μια θα έχουμε μία καλή μεταρρύθμιση και από την άλλη μεριά μία καλή διαρθρωτική πολιτική με έναν προγραμματισμό εξάντια. Τώρα, εμείς θα πρέπει να ερμηνεύουμε τις δεσμεύσεις των κρατών μελών, ό,τι ανέλαβαν τα κράτη-μελή στα πλαίσια του Συμφώνου Ανάπτυξης. Όλα αυτά πρέπει να τα ερμηνεύσουμε στην πράξη μακροπρόθεσμα και θα καταθέσουμε τροπολογίες σχετικά και ελπίζουμε ότι έτσι θα έχουμε μια καλή λύση. Ευχαριστώ Ζανπόλ. Ο Ζομπόλ. Εγώ δεν θέλω να μονοπολίσω το λόγο, θέλω απλώς να σημειώσετε ότι στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών θα πρέπει να οργανωθούμε για το χρόνο ομιλίας αυτού του είδους συζητήσεων, όπου ο καθένας τελικά αισθάνεται άσχημα έστω και αν έχει χρόνο ομιλίας. Βεβαίω, συμφωνώ. Δυστυχώ δεν έχουμε αρκετό χρόνο συνεδρία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Συμφωνώ πάντω. Έχουμε λίγο χρόνο σε σχέση με το φόρτο εργασία. Η Σοφή, η επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να μην υπερβώ το χρόνο μου. Ε, καλωσορίζω το σχέδιο έκθεση κυρια Τάισεν και μπορώ σχετικά εύκολα να εστερνιστώ και όσα είπε και οι τροπολογίες μας ε, θα ευθυγραμμίζονται με αυτήν, θα ενισχύουν περισσότερο τις ε, διάφορες ε, απόψεις της έκθεσης παρά θα τις αποδυναμώνουν. Και όπως είπατε, το Συμβούλιο έχει την τάση να κάνει τολμηρές δηλώσεις, ε, μεγαλεπίβολες υποσχέσεις και προτάσεις και την επόμενη μέρα να παλιδρομούν και να υπαραχωρούν. Λάθος μήνυμα δίνουν προς τους Ευρωπαίους πολίτες. και είναι λάθος μήνυμα και προς τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί φαίνεται να ομφαλοσκοπούμε και να ενδιαφερόμαστε περισσότερο τι συμβαίνει με εμά παρά τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν το ευρύτερο πλαίσιο. Όντω τα πράγματα προχωρούν με ηλικιώδη ταχύτητα και προσοχή να αποφύγουμε να επαναλαμβάνουμε τις μάχες του παρελθόντος, να είναι σαφής η κατεύθυνσή μας. Γιατί ακόμη ε, και αν θέλουμε να υπάρχει ο κόσμος, στον κόσμο ένα κουμπί που να πατάμε και να σταματάει ο χρόνος, δυστυχώς τέτοιο δεν υπάρχει. Ο κόσμος προχωράει με τη δική του ταχύτητα, οπότε τα ημίμετρα, τα ευαλωματικά μέτρα, όλα αυτά είναι παροχημένα και αναποτελεσματικά. Και οι προτάσεις κυρία Τάισεν ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Τα προβλήματα που έχουμε σήμερα δεν ε, είναι απόρρια της ε, ε, ραγδαίας ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αντίθετα της αργής της ε, εξέλιξης. Και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι στιγμής έχουμε διευκολύνει τα πράγματα ε, και έχουμε καταλήξει σε πολλές λύσεις, αλλά θα πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε, γιατί μερικές φορές και εμείς φρενάρουμε τη διαδικασία και θα το τροχοπέδι. Τώρα, για τη δημοκρατική νομοποίηση. Δημοκρατική νομοποίηση δεν σημαίνει μόνο λογοδοσία των θεσμικών οργάνων. Είναι ένα σύστημα που ε, δημιουργούμε και που εξαρτάται και από την όλη διαδικασία που μας οδηγεί στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ας μην ξεχνούμε ότι χρειαζόμαστε την υποστήριξη του κόσμου. Δεν έχουμε εδώ μόνο ε, κάποιες συσκέψεις ε, σοφών ε, που γίνονται και κλεισμένων των θυρών και κάνουν τις συμφωνίες μεταξύ τους. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια πραγματική πολιτική ένωση, είναι ένα τμήμα της ε, συνολικής λύσης. Σε ό,τι αφορά τις α, ε, ε, λεπτομέρειες για την ανάθεση της εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σωστά η συγγετρία λέει ότι εδώ έχουμε διάφορα διλήμματα ως προς την ανεξαρτησία της έκτη, για παράδειγμα. Το γεγονός ότι δεν καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη, Φερρυπίν. Και ταυτόχρονα θέλουμε και οφείλουμε να προχωρήσουμε γοργά και να αναζητήσουμε ρεαλιστικές λύσεις. Πάντως, ό,τι και να κάνουμε, πρέπει να μεριμνήσουμε ότι τα εποπτικά, ε, το εποπτικό έργο θα διαχωρίζεται σαφώς από, τα, από τις υπόλοιπε δραστηριότητες και να καλύπτονται και οι χώρες εκτός Ευρωζώνης, γιατί και αυτές οι χώρες έχουν περισσότερες τουλάχιστον βλέψεις να μπουν κάποια στιγμή στην Ευρωζώνη. Επίσης, είμαι υπέρ μιας πλήρους τραπεζικής Ένωσης που θα έχει τρεις πυλώνες και όχι μόνο την εποπτεία και ταυτόχρονα δεν μπορούμε να φτιάχνουμε ένα πόδι, ένα πυλώνα και μετά να αφήνουμε τους υπόλοιπους δύο για το μέλλον. Και συμφωνώ σε ό,τι αφορά την αμοιβαία, τον επιμερισμό ή την αμοιβαία ανάληψη του δημόσιου χρέους, συμφωνώ με αυτά που λες επίσης ε, για την δημιουργία της θέσης του Υπουργού Οικονομικών. Είμαστε υπέρ και ένας τέτοιος υπουργό, επίτροπος, δεν ξέρω πώς θα λέγεται, θα πρέπει να είναι και προσωπικά υπόλογος. Γιατί αυτό, αυτή είναι μία από τις αδυναμίες του συστήματος. Έχουμε μόνο συλλογική λογοδοσία και συλλογική ευθύνη. Υπάρχει και ατομική. Επίσης, ε, στην έκθεση λέμε μια ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση. Φαίνεται όμως να επικεντρωνόμαστε στο, νομισματικό σκέλος. Να μην ξεχνούμε και το οικονομικό σκέλος. Εσωτερική αγορά, έχουμε πολλές συστάσεις ε, στην Ευρώπη 2020, καινοτομία, αγορά εργασία, συντάξεις και το καθεξής. Ευχαριστώ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, Σόφη. Φαίνεται όμως πως έχει σειρά. ο Φίλιπ. Καλά, Φίλιπ. Αλλάξατε σειρά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Μαριάν, για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι Λυπάμαι, δεν συμφωνώ μαζί σας με το ότι πρώτον μπορούμε να λύσουμε την κρίση μόνο με τα όργανα που διαθέτουμε με βάση τις ισχύουσες συνθήκες και δεύτερον ότι νομικά δεν μπορούμε να πάμε πέρα από αυτές. Τι γίνεται πολιτικά αυτόν τον καιρό. Ο Χέρμαν Βαν Ρόμποϊ αργά και σταθερά και συνειδητά ε, ξεπερνά τις συνθήκες. Τώρα όμως έχουμε την έκθεση, τη νέα έκθεση η οποία ξεπερνά τη συνθήκη και εδώ εμείς στο κοινοβούλιο το κοιτάμε έτσι λίγο φοβισμένοι, προσεκτικά, ενώ εμείς θα έπρεπε να είμαστε αυτοί που σκέφτονται παραπέρα. Το Συμβούλιο δείχνει περισσότερη, περισσότερες ε, αρχικικές ικανότητες από ότι εμάς, ηγετικές ικανότητες. Όπως και στην έκθεση για τα ευρωομόλογα. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε με τις ισχύουσε συνθήκες και τι μπορούμε να κάνουμε πέρα από αυτές τις συνθήκες. Δεν νομίζω πως πρέπει να διστάζουμε να προχωρήσουμε πέρα από τις συνθήκες, ιδιαίτερα σε αυτό που είπα και χθε, πιστεύω ότι σε μια τραπεζική ένωση είναι άσκοπο να κάνουμε λίγο γι' αυτό, γιατί φυσικά όλες οι θέσεις θα καθοριστούν από την ε, νομοθετική έκθεση. Όσον αφορά την νομισματική ένωση, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορούμε να προσθέσουμε. Και να συμφωνήσω με αυτό που είπε η Σόφη για την Ευρώπη 2020. Πολλοί το ξεχνούν. Επιμένουμε να κάνουμε αυτές τις δεσμεύσεις όσο το δυνατόν περισσότερο δεσμευτικές γίνεται. Το εννοούμε ή όχι. Ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης πρέπει να, να θέσουμε αυτή την προτεραιότητα ακόμα πιο πάνω. Πρέπει πραγματικά να ε, μονιμοποιήσουμε την ισχύ των, ε, αυτών των έκτακτων ε, συνθήκων. Επίσης, το θέμα της λογοδοσίας. Ο Λίαμ είπε ότι δεν θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα ούτε στις ε, περιφερειακές χώρες, ούτε στις ε, κεντρικές, ούτε στους ε, δότες, ούτε στους ε, Δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε τίποτα χωρίς αυξημένη λογοδοσία. Και χω, χωρίς τη λογοδοσία δεν γίνεται τίποτα. Ακόμα και με την κατάσταση που έχουμε σήμερα δεν είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσουμε να τους πείσουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα από αυτά που έλεγε ο κύριος Βεστέρ Εάν, εφόσον Εάν το κοινοβούλιο δεν μπορεί να πιέσει για αύξηση της λογοδοσίας, δεν ξέρω ποιο, ποιο είναι το έργο μας εδώ πέρα. Η δημοσιονομική αλληλεγγύη είναι το σημαντικότερο, το κυριότερο. Εάν θέλετε εάν θέλετε να ξεπεράσουμε την κρίση, να προωθήσουμε τη δημοκρατία, χρειάζεται αυτή η αλληλεγγύη. Εάν είναι ένα πράγμα το οποίο θα αφήσουμε στις επόμενες ε, γενιές είναι η, σωστή δημοκρατική αρχιτεκτονική μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης και όχι μια ομοσπονδία τεχνοκρατών που δεν θα είναι αρεστή σε κανέναν. Εγώ είμαι δημοκράτης πρώτα απ' όλα πριν την ιδιότητα του πράσινου, πριν την ιδιότητα του Ευρωπαίου. Είμαι δημοκράτης και αυτό πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητά μας ως πολιτική. Και πραγματικά θα ήθελα να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό και να μην επαναλάβουμε σε αυτή την έκθεση αυτά που έχουν ήδη υποθεί. Μαριάννα, λοιπόν... Ξέρω ότι προσπαθήστε να κάνετε ένα σπαγκάτο ουσιαστικά και εξού και η μεγάλη διαφορά μεταξύ της ε, αρχικής έκθεσης και της, ε, του σχεδίου που υποβάλλατε τώρα. Πραγματικά όμως ήσταν πολύ στεναρή και καταλήξατε σε ένα πολύ αξιόλογο έγγραφο. Ευχαριστώ. Ο Ήβο. No tak, tak když jsem tak poslouchal Filipa, tak... Ακούγοντας τον Φιλίπ, κατάλαβα γιατί ο Ζαν Πολ Γκοζές είπε να μην ε, αισθανόμαστε τόσο καταπιεσμένοι κατά αυτές τις συζητήσεις. Τώρα όμως το καταλαβαίνω. Και εγώ θέλω να ορίσω εκ μέρους της ομάδας μου το γενικό προσανατολισμό των τροπολογιών. Καταρχήν το πλαίσιο. Στο εκτιμώντας ε, δέλτα είναι πολύ πιστικό. Σε ένα παράδειγμα, όπου θα έχουμε είτε μια συγκεντρωτική Ευρώπη, η οποία θα αντιμετωπίζει παθητικά τις εξελίξεις του κόσμου. Αυτό όμως εμείς δεν το θέλουμε. Εμείς πρέπει να πούμε ότι η αλήθεια στην οικονομία είναι η υπόθεση των μονοπωλίων. Η έκθεση ορίζει μία χαμηλή δυνατότητα ανάπτυξη, σημαντικό έλλειμμα και γενικά κρίση. Μπορούμε να το βάλουμε αυτό, αλλά εγώ πιστεύω ότι πουθενά στην έκθεση δεν γίνεται μια ακριβής συζήτηση για τις αιτίες... Μπορούμε να έχουμε μία διαφορετική ιδέα για το ποια είναι η αιτία, αλλά η έκθεση δεν λέει τίποτα. Για μας είναι απαράδεκτο να χωρίζουμε την Ευρώπη σε ε, Ευρώπη των κεντρικών χωρών και των περιφερειακών χωρών. Εάν εμείς πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια για την οικονομική ένωση της Ευρώπης, Μία τέτοια διάκριση οδηγεί σε αποτυχία αυτών των συζητήσεων. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, όποιο είναι στο κέντρο πάντα έχει δίκιο, έχει δίκιο και όποιος είναι στην περιφέρεια πάντα έχει άδικο. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό η σημερινή, αυτή η διαδικασία η οποία θα πρέπει να τελειώνει με ομοσπονδιοποίηση Θα έπρεπε λοιπόν αυτή η διαδικασία να την χάνει σοβαρού ελέγχου. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, χρειάζεται συζήτηση με τους πολίτες, με τα εθνικά κοινοβούλια. Η διαδικασία επικύρωσης που απαιτεί την τροποποίηση των συνθήκων θα πρέπει να είναι συμβατή με τις συνταγματικές ανάγκες και ισχύοντα των κρατών μελών γιατί άμα δεν έχουμε αυτή τη βάση είναι άτοπο να συζητάμε για την επιτυχία αυτού του σχεδίου στο μέλλον. Στη συνέχεια, ο ενιαίος μηχανισμός εποπτείας Σε αυτήν την ομάδα έχουμε περισσότερο κόσμο, ο οποίος έρχεται από χώρες που δεν είναι στην Ευρωζώνη αλλά θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη της εμπροζώνης θα ήθελαν τα δημοσιονομικά τους ιδρύματα να υπόκεινται σε ένα νέο σύστημα εποπτείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όμως ποιος θα έχει τα τη τελευταία λέξη, τα κράτη-μέλη που δεν είναι μέλη της εμπροζώνης και έχουν απλώς τράπεζες που λειτουργούν στην επικράτειά τους και ανήκουν σε μητρικές τράπεζες οι οποίες ε, ε, ε, ανήκουν σε χώρες που ανήκουν στην Ευρωζώνη. Εγώ είμαι Τσέχος. Η κεντρική μου τράπεζα ασκεί εποπτεία στις τράπεζες. Αλλά τι γίνεται όταν ξεπερνά αυτά τα όρια, για την εγγύηση των καταθέσεων, όταν ε, το επιτόκιο, το εξωτερικό επιτόκιο είναι πάνω από το εθνικό επιτόκιο, δηλαδή δεν υποσκάπτεται έτσι η δημοσιονομική ανεξαρτησία ενός κράτους μέλους και η παρουσία δύο κατηγοριών τραπεζών, μία που θα έχει άμεση πρόσβαση στα δημόσια, ε, ε, ε, στα δημόσια κονδύλια και μία όχι. Και αυτό για μας είναι απαράδεκτο. Και αυτό που λέγεται επίσης για την φορολογική εναρμόνιση είναι απαράδεκτο για μας. Μαρίσα τώρα από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτριά μας, γιατί πραγματικά μας έδωσε μια εξαιρετική βάση εργασίας. Μια και έχω λίγο χρόνο, θα περάσω κατευθείαν στο ψαχνό, στα πιο επίμαχα θέματα της έκθεσης. Όντως, ε, είχαμε κάποια πρόοδο στις εργασίες, γιατί για να είμαι ειλικρινής, το, η αρχική πρόταση του Συμβουλίου και του Πρόεδρου Βαν Ρόμποϊ με τίτλο «Προς μία γνήσια οικονομική και νομισματική ένωση». Ε, αφενός όμως ε, η συντάση με τέτοια έκθεση αφετέρου εγκαταλείπει στη μοίρα του χώρα του Νότου είναι η έκθεση αυτή του κυρίου Βαν σαν παραπλανητική διαφήμιση θα πρέπει να συζητήσουμε πραγματικά να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στην πρόταση αυτή. Μία από τις προτάσεις είναι η μνήμα της ανάγκης επίδειξης αλληλεγγύης προς τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Συμφωνώ, αλλά δεν, δεν συμφωνώ με την αιρεσιμότητα, με τους όρους που συνοδεύουν ε, αυτή την αλληλεγγύη. Γιατί ουσιαστικά ε, τροφοδοτούμε την λογική της απόκλησης, της διαφοράς και της ε, de facto ανισότητας που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων χωρών της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Επίσης, ήθελα να επαναλάβω αυτό που λέει η συγκήτρια. Θα πρέπει να χαράξουμε το δρόμο προς την κοινή ανάληψη χρέους. Διαφωνώ και πάλι όμως με τους όρους που επισυνάπτονται σε αυτή την ανάγκη. Γιατί λέμε να θέσουμε αυστηρές προϋποθέσεις ώστε να αποφύγουμε εσπευσμένη δράση. Αλλά αν δούμε τους όρους, όπως είναι η, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και πολλούς όρους, μεταρρυθμίσεις, δημοσιονομικές πειθαρχίες, ένα σύνολο όρων που συνοδεύουν αυτή την πρόταση, που είναι δύσκολο να τηρηθούν. Το θέμα δεν είναι ότι δεσπεύδουμε, αλλά ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να εκπληρώσουμε όλε αυτέ τις προποθέσει για να καταλήξουμε σε κοινή ανάληψη χρέους ή κοινό χρέο. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε κατάματα αυτή την πραγματικότητα, αν θέλουμε πραγματικά να εμφανθύνουμε. Δεν μπορούμε να περιορίζουμε περιορίζουμε σε αναγγελίες αγαθών προθέσεων. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και αν πραγματικά θέλουμε κοινό χρέος, κοινή ανάληψη χρέους, να δούμε πώς θα το καταφέρουμε. Και δεν είναι μόνο θέμα ότι να αποφύγουμε τη σπουδή και την εσπευσμένη δράση. Ένα άλλο θέμα. Ενίσχυση του δημοκρατικού ελέγχου. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον ολοκληρωμένο μηχανισμό υποπτία τη ΕΚΤ. Ποιο είναι ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενισχυθούν γενικώ ε, οι διάφορε μορφέ δημοκρατικού ελέγχου, αλλά αυτή η αιμονή στην διατήρηση τη ανεξαρτησία τη ΕΚΤ. Ό,τι ενίσχυση με την ενίσχυση που αποκτά η παρουσία της ΕΚΤ και με τις απαντήσεις που έδωσε στην κρίση, δεν έχουμε καμία δυνατότητα για αξιόπιστη λογοδοσία εκ μέρους της ΕΚΤ, γιατί έχουμε μια πραγματικά αδιάλακτη και κλειστή λογική ως προς την ανεξαρτησία της ΕΚΤ, που δεν μας βοηθάει να επιλύσουμε τα προβλήματά μας. Επίσης, προσπαθώντας να ενισχύσουμε τη δημοκρατική νομοποίηση, το ρόλο του δημοκρατικού ελέγχου. Θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι και να διακόψουμε μια πολύ κοινή τάση πολλών εγγράφων που μελετήσαμε και που είναι η τάση να δημιουργούμε πληθώρα μηχανισμών, συμφώνων, οντοτήτων, ενιών. Πολλαπλασιάζουμε τις διάφορες μας αντιδράσεις χωρίς όμως κανέναν δημοκρατικό έλεγχο όλων αυτών των νέων εργαλείων, μηχανισμών, συστημάτων, συμφώνων, προβλημάτων, αρχών, οργανισμών, οντοτήτων. Δεν έχουμε δημοκρατικό έλεγχο όλων αυτών. Και απομακρύνουμε όλο και περισσότερο τους συμπολίτε μας από την οποιαδήποτε συμμετοχή σε λήψη απόφασης για όλα αυτά τα κατακαιρματισμένα μας μέτρα. Δεν μπήκαμε καν στον κόπο να κάνουμε μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των συνεπειών αυτού του ακατάσχετου πολλαπλασιασμού των ε, μηχανισμών. Ενώ λείπει το ουσιώδες, που είναι ο δημοκρατικός έλεγχος, η δημοκρατική νομιμοποίηση για να επέμβουμε και να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Έχω λοιπόν διάφορα σχόλια, αλλά σε αυτά τα σημεία κυρίως ε, απομακρυνόμαστε κάπως από τη θέση της αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε και περαιτέρω. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους όσους ε, τηρούν ευλαβικά το χρόνο τους. Θα δώσω το λόγο και στον κύριο Γκουαλτιέρη που έχει πολλαπλές ιδιότητες. Είναι αναπληρωτής ε, στην ΕΚΟΝ, είναι εισηγητής ε, της έκθεσης στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και είναι και στην ομάδα των αρμόδιων κομματικής πειθαρχία του ΕΛΚ. Ρομπέρτο Γαλτιέρη. Λοιπόν, το κείμενό μου είναι έτοιμο. Εγώ εδώ θα, θα σας δώσω τα εννέα κεντρικά σημεία. Είναι συμβατή με τη θέση της έκθεσης της Μαρίας Τάισεν, την οποία ευχαριστώ για τη συνεργασία και θέλει να την ενισχύσει από ε, συνταγματικής πλευράς. Το πρώτο αφορά στις αλλαγές. Σίγουρα μία ουσιαστική αλλαγή των συνθήκων χρειάζεται για σταθερότητα, να προσδώσει σταθερότητα στην νομισματική ένωση. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασκήσει πλήρως τις θεσμικές του αρμοδιότητες στα πλαίσια της, του δικαιώματος πρω, πρωτοβουλίας για την μεταρρύθμιση των συνθήκων. Δεν μπορούμε να έχουμε εμείς μία συνδιάσκεψη πριν από το 2015. Δεν είναι καν χρήσιμο. Μία διαδικασία η οποία, την, την οποία την αφήνουμε μόνο στα χέρια των, θε, θεσμικών τεχνικών ε, είναι κάτι το οποίο δεν θα συμμερίζονται μετά οι πολίτες. Συμφωνώ λοιπόν με αυτό που λέει η έκθεση Τάισεν, ότι, η, ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μία μεταρρύθμιση των συνθήκων το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προετοιμάσει αυτήν τη μεταρρύθμιση και δεν θα πρέπει αυτό όμως να μας εμποδίζει να δράσουμε ίσα ίσα, πρέπει να δράσουμε γρήγορα μέσα στο νομικό πλαίσιο των συνθήκων που επιτρέπουν πρώτον να προχωρήσουμε πολύ πιο μακριά από ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και δεύτερον επιτρέπουν ε, και προβλέπουν μία πολυεπίπεδη governance για μία πιο στενή ολοκλήρωση των χωρών εκείνων που θέλουν να, ε, να ενωθούν παραπάνω, πόσο μάλλον εκείνων που έχουν το ίδιο νόμισμα. Α, από συνταγματικής πλευράς η Τραπεζική Ένωση θα πρέπει να μπει σταθερά και αμετάκλητας μέσα σε ένα γενικότερο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα δυναμίας της οικονομικής διακυβέρνησης. Πρόκειται για έλλειψη δημοκρατικού ελλείμματος. Πρόκειται για την απονομιμοποίηση εκ μέρους των πολιτικς του κεντρικού οργάνου. Αυτό εμείς μπορούμε να το ξεπεράσουμε ενισχύοντας τον κατάλογο των θεσμών που έχουμε στη διάθεσή μας, όχι να δημιουργήσουμε νέα όργανα εκτός ένωσης. Για τα τέσσερα μπλόκα τώρα. Από συνταγματικής πλευράς έχουμε λίγα πράγματα να πούμε, δεν λέμε τίποτα. Θυμίζουμε μόνο ότι οι συνθήκες επιτρέπουν τη διαδικασία της πασαρέλας που επιτρέπουν να μεταρρυθμίσουμε μια ειδική νομοθετική διαδικασία σε τακτική νομοθετική διαδικασία. Για την φορολογική ένωση το πρώτο σημείο είναι να υπογραμμίσουμε και από θεσμικής πλευράς την αδυναμία να ενισχύσουμε την governance του ευρώ μέσα στα πλαίσια ενός μοντέλου ένωσης κανόνων. Θα πρέπει να έχουν Ένωση και η Ευρωζώνη μία δική της φορολογική δυνατότητα και έχουμε και διαδικασίες που μπορούν να μας επιτρέψουν να αναπτύξουμε αυτές τις εξελίξεις και μέσα στο τωρινό πλαίσιο ε, θα μπορούσαμε να έχουμε το θέμα της καταβολής στην ε, Ευρωζώνη και μετά στην ε, γνώμη ορίζουμε με δρόμους ούτως ώστε αυτό το τόσο σημαντικό μέτρο να ενταχθεί μέσα στις εσωτερικές διαδικασίες προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι αν διατρέχουμε το συγκεκριμένο κίνδυνο να έχουμε έναν εξωτερικό διακυβερνητικό υπολογισμό της Ένωσης και αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Από φορολογικής πλευράς λέμε ότι το άρθρο 136 θα μας επέτρεπε να προχωρήσουμε και πέρα από αυτά τα οποία έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Έχουμε το, να δούμε το συντονισμό και την επίπεδη εποπτεία. Πρέπει να ενισχύσουμε και το ρόλο του Κοινοβουλίου και υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις. Η άλλη θέση αφορά στο μηχανισμό σταθερότητας, συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, όπου αναφέρουμε, δίνουμε εδώ έναν μηχανισμό περίπου αποφασιστικό, αποφασιστικό δυνατότητας, όμως τέλειωσα το χρόνο μου και θα σας δώσω το γραπτό. Συγγνώμη, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε, αλλά έχουμε πολλούς ομιλητές. Τώρα περνάμε στο τρίλεπτο αναομιλητή. Ο Βέρνερ. Ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ τις απόψεις της ησυχητρίας όμως διαφωνώ πλήρως με την έκθεση. Υπάρχουν 35 αναφορές σε ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, 100 αιτιολογικές σκέψεις και 5 ε, αιτήσει στην σελίδα 17 και παραρτήματα τα οποία αναφέρονται στην νομοθεσία και είναι και αυτά πολυσέλιδα. Πιστεύω πως ούτε πολιτικά ούτε και λογικά είναι αυτό εύκολο να εφαρμοστεί. Γι' αυτό σας παρακαλώ να συγκεντρωθείτε σε αυτό που εμείς ζητούμε. Και ποιο είναι αυτό? Στην σελίδα 17 η Κομισιόν ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συνομοθέτη κτλ. κτλ, κτλ να, συγκατα... να δώσει τη, συμφωνή... τη συγκατάθεσή του ναι. Τότε πρέπει ο και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι και αυτός ο μέλος, ένας από τους πέντε που βρίσκονται στο Προεδρείο που ασχολείται με αυτά. Πρέπει να συμμετέχουμε και πιο ενεργά ως συνομοθέτης. Και εκτός από αυτό πρέπει να προσέξουμε, να αποφύγουμε τον κίνδυνο με σκοπό να δημιουργήσουμε μια καλύτερη τραπεζική εποπτεία, να χωρίσουμε την Ευρώπη, να την διχάσουμε. Ο κύριος Ρομπόη την πρώτη ε, θέση του στις 26 ε, Ιουνίου είπε εποπτεία με ανάμιξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και είναι τελείως διαφορετικό αυτό από αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Κανένας δεν πρέπει να διχάσει την Ευρώπη προσπαθώντας να ενώσει τα τραπεζικά συστήματα. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Κοιτάξτε εδώ. Τα πιο σημαντικά τα χάνουμε και αναλώνουμε χώρο και χαρτί με περιτά, περιτές αναφορές. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σας καλώ να συγκεντρωθούμε στο ουσιώδες και να δούμε τι θέλουμε. Θέλουμε να εργαστούμε παράλληλα, μαζί. Φυσικά και το θέλουμε. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και να ενισχύσουμε τα δημοκρατικά μας δικαιώματα. Φυσικά ο κύριος Φερχόφστας, ο Κον Μπέντιτ, ο, ο πρόεδρος, ο κύριος ε, Σούλτς, ο Έλμαρ Μπρόκ, είναι, εκείνοι που, θέλουν να συνοδεύσουν το έγγραφο του Χερμάνου Βαν Ρόμποϊ. Και τι κάνουμε εμείς, χάνουμε την ουσία με τις τροπολογίες. 110 είναι αυτές. Και πραγματικά σας παρακαλώ να μην χάνουμε έτσι την ουσία, να πάρετε τα πράγματα στα σοβαρά και να κάνουμε μία ουσιώδης πρόταση δύο σελίδων που να αποκρισταλώσει τις συζητήσεις μας σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να υπερασπίσω την εισηγήτρια σε ό,τι αφορά τη μορφή της έκθεσης, γιατί ε, είμαστε δεσμευμένοι να χρησιμοποιούμε αυτή τη μορφή όταν έχουμε εκθέσεις πρωτοβουλίες νομοθετικές. Πρέπει να έχουμε τόσο τέτοιες αιτιολογικές εκθέσεις ε, μετά το, το διατακτικό και το παράρτημα. Τα παράπονά σας στη διάσκεψη Προέδρων, αλλάξει τους κανόνες, αν διαφωνείτε. Λυπάμαι, Βέρνερ, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω. Πίτερ Σέιμον. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Φυσικά, είναι σημαντικό αυτό που είπαν οι συνάδελφοι να αναλάβουμε πρωτοβουλία. Πρέπει όμω να παραμείνουμε σοβαροί, να διατηρήσουμε στη σοβαρότητά μα, γιατί όταν οι άλλοι δεν είναι, πρέπει να έχουμε εμεί το έργο να επαναφέρουμε τη συζήτηση στι ράγες και να δούμε πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα καλύτερα στοιχεία χωρί να υποστούμε τι συνέπειε των πιο άσχημων στοιχείων. Χρειαζόμαστε μια ενιαία, ένα ενιαίο ε, σύστημα εποπτείας και ασφάλειας στην Ευρώπη. Αλλά Πώ θα γίνει αυτό, Αυτό θα γίνει με συγκεκριμένε προποθέσει, με τι κατάλληλε προποθέσει, όχι έτσι όπω είναι τώρα. Και όσο ε, στα πλαίσια τη εποπτεία δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν οι τράπεζε αξιολογούνται με τον ίδιο τρόπο, τότε πώ μπορούμε να αγγιθούμε στου επενδυτέ ότι τα δικά του χρήματα, οι δικέ του ε, αποταμιεύσει είναι ασφαλείς. Όσο παραμένουμε στα λόγια και στις ε, συζητήσεις δεν γίνεται τίποτα. Όσο το κοινοβούλιο δεν είναι αναμεμειγμένο στο, στο έπακρο, τότε δεν μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό. Η Κομισιόν και το Συμβούλιο μας μιλάνε για, για συστημικούς ε, ελέγχους, για τραπεζικές εποπτείες, όμως κινδυνεύουμε να επέλθουμε σε μια πολύ άσχημη κατάσταση, σε μια πολύ άσχημη εποπτεία, η οποία θα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε μια πολύ μεγάλη κεντρική ευρωπαϊκή τραπεζά, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την εξυγίανση όλων των υπολείπων. Και αυτό, αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση καλό. Αυτό βλάπτει και τους επενδυτές και τις επιμέρους τράπεζες. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά, που χρήζουν διευκρίνησης. Και αυτά τα ερωτήματα δεν θα απαντηθούν μόνο και μόνο βάζοντας όλες τις τράπεζες μαζί υπό μία μητέρα εποπτική τράπεζα. Και θέλω να ρωτήσω πώς μπορούμε να εργαστούμε για τη δημιουργία ενός, ε, ενός ε, οργάνου το οποίο θα φροντίζει για την σωστή εποπτεία χωρίς να κάνει κατάχρηση εξουσιών, το οποίο θα εγγύεται στους επενδυτές και στους καταθέτες την ασφάλεια των καταθέσεών τους, το οποίο θα ασχολείται όχι μόνο με το σύνολο αλλά και με τα επιμέρους συστατικά στοιχεία, το οποίο δεν θα βάζει σε κίνδυνο τους καταθέτες. Εάν δεν μπορεί αυτό να το εξηγήσει συνολικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει να θέσουμε ξεκάθαρες προϋποθέσεις, κάτι που προς το παρόν δεν συμβαίνει. Και πραγματικά περιμένω από όλες τις ομάδες να συνεργαστούμε καλά και να θέσουμε τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες θα δημιουργήσουμε ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα σε όλα τα κράτη-μέλη και στο τέλος της ημέρας η πρόεδρος Πίτερ με συγχωρείς, έχει ξεπεράσει το χρονικό όριο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, 15 λεπτά πριν ε, ολοκληρωθεί ο χρόνος σας, θα σας προειδοποιώ με το σφύρι. Νέα μέθοδος. Η Ελίζα. Ευχαριστώ. Σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η Μαριάν ε, επιτέλεσε ένα πολύ αξιόλογο και πολύ μεστό έργο. Σε ό,τι αφορά την έκθεση του Βαν Ρομπόι, Ας μην ξεχνούμε τους τέσσερις άξονες. Ως προς τον πρώτο άξονα, η θέση της Μαριάννα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Και σε τελική ανάλυση καλύπτει η πρόταση αυτή του, της χρηματαγορές και αυτό που λέμε τραπεζική ένωση. Οπότε ας αφήσουμε τον πρώτο άξονα, ας δούμε τους άλλους τρεις άξονες. Εκεί μιλάει για ένα μέσο και μάκρο πρόθεσμο όραμα ο Βαν Ρομπέη. Αλλά εκεί δεν λαμβάνει ε, αρκετά υπόψη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τη Δημοσιονομική και την Οικονομική Ένωση. Για τη Δημοσιονομική Ένωση η Μαριάν μα υπενθυμίζει ένα τμήμα του διπλού πακέτου, αλλά ένα μόνο που αφορά τον έλεγχο στου εθνικού προπολογισμού. Ξέχασε όμω τα βήματα που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την διαχείριση του δημοσίου χρέου. Έχουμε πολλά έγγραφα και ήδη έχουμε καταλήξει συνένεση. Τώρα θα πρέπει να διατρανώσουμε τη θέση μας απέναντι στις στα άλλα θεσμικά όργανα. Ε, μιλήσαμε για τα, το δημόσιο χρέος, την αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους, για τα ομόλογα σταθερότητα πριν το, το εξαπλό πακέτο. Τώρα έχουμε το διπλό πακέτο και το συναφές χρονοδιάγραμμα. Δημοσιονομική ένωση δεν σημαίνει μόνο έλεγχος επί των προϋπολογισμών. Επίσης, θα πρέπει τα μηνύματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να περιληφθούν στην έκθεση αυτή. Για παράδειγμα, στη συζήτηση για τους ε, ιδίους πόρους ή το φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Και για αυτά τα θέματα έχουμε δεδηλωμένες θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα πρέπει να τις διατρανώσουμε. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται η Δημοσιονομική Ένωση. Αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να ενισχυθεί. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά την Οικονομική Ένωση. Η έκθεση του Ρομπέη επισημαίνει τις ανισορροπίες που υπάρχουν στην Ένωση και θεωρεί ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά δεν λέει και τίποτα ουσιαστικό εμείς θα πρέπει να προτείνουμε κάτι ουσιαστικό. Και στο διπλό πακέτο αναφέρεται 1% του ΑΕΠ να δοθεί σε αντικυκλικά μέτρα, να δημιουργηθεί η στρατηγική για την απασχόληση, γιατί σε επισκόπηση ανάπτυξης, η Ευρώπη 2020. Να πούμε και εμείς τις, γνώ... τις απόψεις μας για τα θέματα αυτά, αυτό το κεφάλαιο. Και κάτι άλλο. Για τα τέσσερα κεφάλαια, για τους τέσσερις άξονες που προβλέπετε, αρκούν αυτά ή να προσθέσουμε και ένα πέμπτο για τις κοινωνικές συνθήκες και για το κράτος πρόνοιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί γιατί θα πρέπει να αρκεστούμε στην κατάρρευση του κράτους πρόνοιας και της ευημερίας των Ευρωπαίων πολιτών, γιατί σε αυτή την, και σε αυτή την κοινωνική ευημερία στηρίζεται η δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα. Ευχαριστώ. Η Αστρίδη Λούλινγκ. Εγώ θα ήθελα να κάνω δύο σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτη, αναρωτιέμαι για τη χρήση αυτής της έκθεσης πρωτοβουλίας για τη χρησιμότητα αυτής της έκθεσης πρωτοβουλίας αφού έχουν ήδη παρουσιαστεί μέρη των κειμένων σχετικά με την Τραπεζική Ένωση. Αναρωτιέμαι λοιπόν μήπως ε, εδώ απλώς ε, κάνουμε μία άσκηση στυλ. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε τις επικαλύψεις, διότι ήδη βιαζόμαστε. για να γνωμοδοτήσουμε επί των νομοθετικών προτάσεων. Γιατί λοιπόν να χάνουμε χρόνο, τον οποίο δεν έχουμε με μία έκθεση πρωτοβουλίας ε, που σε μεγάλο βαθμό ασχολείται ακριβώς το ίδιο θέμα. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Και μία δεύτερη παρατήρηση, πιο ουσιαστική, σχετικά με την Ένωση των Τραπεζών που είναι απαραίτητη. Βρισκόμαστε σε μία δυσεπίλητη εξίσωση. Από τη μια θα πρέπει να προστατεύσουμε την ενιαία χρηματοπιστωτική αγορά της Ευρώπης των 27 και από την άλλη μεριά η κρίση του ευρώ προχωράει. Όλοι όσοι δεν βρίσκονται στην ευρωζώνη θα το θελήσουν ή μπορεί και να μην μπορέσουν να συμμετέχουν. Η Ευρωζώνη πρέπει να προχωρήσει μακρύτερα στην ολοκλήρωση για να επιβιώσει μεσοπρόθεσμα. Αυτό όμως ε, θα οδηγούσε σε έναν κατακαιρματισμό της ενιαίας αγορές. Τώρα αν πάρουμε την αντίστροφη θέση είναι σαφές ότι οι χώρες της Ευρωζώνης εξαρτώνται από τις άλλες για την, για την περιφρούρηση του συστήματος. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου και εγώ δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε όλες αυτές τις αντιφάσεις. Πρόκειται για ένα πρόβλημα πάρα πολύ δύσκολο εμείς βέβαια ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, διότι αλλιώς ε, θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Εγώ σταματάω εδώ, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να ξαναγράψουμε μία νέα συνθήκη σε τούτη εδώ την Επιτροπή. Προτεραιότητά μας είναι να μπορέσουμε έγκαιρα να συντάξουμε την έκθεσή μας για τις νομοθετικές προτάσεις που βρίσκονται επιτάπητος. Αυτό θα ήθελε. Σε αυτό πρέπει να συγκεντρωθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος. Σύρπα Πετικάινεν. Ευχαριστώ. Και καλό κουράγιο Μαριάν. Έχεις πολλή δουλειά προσπαθώ να συμφιλιώσεις όλες αυτές τις διστάμενες απόψεις, αλλά πραγματικά δεδομένου του χρόνου που είχες ε, έκανες θαυμάσια δουλειά. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ακόμη πιο πολλοί αριθμές αναφορές ε, στις αποφάσεις που έχει λάβει μέχρι τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία δέκα χρόνια. Και ελπίζω να το περιλάβεις ε, στην έκθεση. Και καλό θα ήταν να φανεί αυτή η συνεπής ε, και συνεκτική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι ισχυρό αυτό το πολιτικό μήνυμα. Τώρα, επίσης, ε, οι κανονισμοί και οι οδηγίες για τις καταχρήσεις αγοράς, για τους οίκους αξιολόγησης, πολλές, ε, πολλά νομοθετήματα για τις χρηματαγορές και τα χρηματοπιστωτικά. Πολύ σημαντικό να αναφερθούν. Ε, βέβαια, έχουμε και την ε, Επιτροπή για την Κρίση, το, την έκθεση για το πακέτο θα τη τα μέτρα εποπτείας, επίσης πολύ σημαντικά. Και σημαντικό θα είναι να λάβουμε υπόψη το χαρακτήρα του πακέτου. Πολλές αποφάσεις θα ληφθούν ως δέσμη μέτρων όχι κάθε πράγμα χωριστά. Αυτή την ιδέα του συνόλου δεν θα πρέπει να την ε, αμελούμε και να την αγνοούμε. Άλλη σημαντική πολιτική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι τα κράτη-μέλη με πολύ κοντόφθαλμο τρόπο αντιμετώπισαν την κατάσταση και με αναποτελεσματικό σε σχέση με τις προσδοκίες και τις ανάγκες των ε, πολιτών. Χρειαζόμαστε μία πανευρωπαϊκή θεώρηση. Συμφωνώ με αναγκαία ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κάνουμε περισσότερα στο ισχύον πλαίσιο, με βάση δηλαδή τις συνθήκες. Και ναι, μεν κάποια στιγμή θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία μεταρρύθμισης των σηκών, αλλά δεν θα πρέπει να είναι αυτό πρόσχημα για να καθυστερήσουμε την ανάληψη δράσης. Το τρίτο πολιτικό μήνυμα είναι αυτό που ανέφερε ο Βέρνερ, να πούμε ότι έχουμε μία Ευρώπη και να αποφύγουμε τις δύο ταχύτητες και δεν θα πρέπει να δημιουργούμε Ευρώπη δύο ταχυτήτων ή δύο διαφορετικά τμήματα στην Ευρώπη, ένα διαχωρισμό. Και όλα τα κείμενά μας αυτό το χαρακτήρα θα πρέπει να έχουν. Επίσης, και η φορολογία θα πρέπει να αποτελεί το του πακέτου και οι αρμοδιότητες για τη φορολογία. Βέβαια, γνωρίζω ότι εδώ είναι κάπως επίμαχο αυτό το θέμα. Και το θέμα το κοινωνικό. Ναι, βλέπω ότι έχω ξεπεράσει το χρόνο μου, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα, σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Το σύστημα εγγύησης καταθέσεων και τα ταμεία για την εξυγίαση των ταμείων. Τα χρήματα θα πρέπει να προέλθουν από τις ίδιες τις τράπεζες και μετά από εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επίση ε, να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος για την τράπεζα και η πόροι σε ό,τι αφορά το μοντέλο για την εξυγίαση. Ευχαριστώ. Δύο ομιλητές μας έχουν απομείνει. Ο Ντιόγκο Φέιο πρώτα. Ευχαριστώ. Καταρχήν, Σάρων, να συγχαρώ θερμά τη Μαριάν Τάισεν για το έργο της υπογραμμίζοντας τη σημασία των δύο εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Και μάλιστα στην έκθεση των τεσσάρων πρόεδρων κρίμα που δεν περιλαμβάνεται και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή είναι η σημαντική μορφή και νομίζω ότι θα πρέπει να τονιστεί στην έκθεση. Ο πρόεδρος του θεσμικού οργάνου που έχει την πιο άμεση σύνδεση με τους πολίτες δεν συμπεριλαμβάνεται σε μια τόσο σημαντική έκθεση των τεσσάρων πρόεδρων. που έχει τίτλο «Προς μία οικονομική και νομισματική ένωση». Για να βρεθούμε στο δρόμο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης θα πρέπει να ασχοληθούμε με, το οικονομικό, με την οικονομική ένωση, με τη δημοσιονομική ένωση, με την τραπεζική ένωση και την πολιτική ένωση. Αυτές είναι οι τέσσερις πτυχές, οι βασικές οι τέσσερις άξονες. Και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασχοληθεί ιδιαίτερα με την ε, σύνδεση της οικονομικής με την πολιτική ένωση. Αυτό λείπει δυστυχώς. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε μια οικονομική ένωση ε, με ένα οικονομικό συμβούλιο που θα συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο ενώ έχουμε ένα ενιαίο νόμισμα. Εκεί θα πρέπει να κάνουμε το ποιοτικό άλμα. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να προσθέσει την ε, συμβολή του και την προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Σε όλες τις ε, ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ασχοληθήκαμε πολλές φορές με τα θέματα αυτά, αλλά νομίζω ότι το μήνυμα που θα πρέπει να προσθέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση είναι ένα σαφές πολιτικό μήνυμα, απερίφραστο πολιτικό μήνυμα. Να δούμε ποιες είναι οι πρόθεσμες προτεραιότητές μας, αλλά ταυτόχρονα με ένα βλέμμα προς το μέλλον. Τι μέλλον θέλουμε για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Δεν μπορούμε να κάνουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση στρέφοντας την πλάτη μας στα κράτη-μέλη. Επίσης, ποια είναι η σχέση των κρατών που βρίσκονται εντός της ζώνης ευρώ και των κρατών που είναι εκτός ευρωζώνης. Πολλά είναι τα θέματα εδώ. Αν δεν λάβει η χώρα μια θεσμική εξέλιξη, πώς θα πλαισιώσουμε τις χώρες που δεν έχουν νέο νόμισμα που δεν έχουν το ευρώ. Θα συμμετέχουν, θα συμμετέχουν και ο θελός, με ποιο τρόπο, πώς θα πλαισιωθούν. Επίσης, το θέμα της δημοκρατικής νομιμοποίησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει ως συνομοθέτη σε πολλά θέματα. Αλλά θα πρέπει να συμμετέχει όλο και περισσότερο σε ένα όργανο ελέγχου των κοινωτικών πολιτικών. Και αυτό είναι ένα θέμα που μας αγγίζει ιδιαίτερα. Και θα πρέπει να το εξηγήσουμε στους πολίτες ότι Αυτά τα πολιτικά ζητήματα είναι θεμελιώδη για να επιληθούν τα υπόλοιπα προβλήματα. Είναι λογική απόρρεια. Νομίζω και αυτό το μήνυμα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις δύο εκθέσεις αυτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Και ο Σβένα τελευταίος. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ την Μαριάν για την έκθεση. Πιστεύω πως είναι σημαντικό να αντιδράσουμε ως κοινοβούλιο με τον ίδιο τόνο ως ε, τη ομάδα του κυρίου Βαν Ρόμποη. Υπάρχουν στην έκθεση Βαν Ρόμποη κάποιες ε, γενικές ε, αναφορές, αλλά εμείς έργο μας είναι τώρα να τις μετατρέψουμε σε κανονικές συστάσεις. Ε, η διατύπωση είναι ένα πρόβλημα και το περιεχόμενο, διότι διαχωρίζονται τα θέματα και γίνεται δυσανάγνωστο και σε αυτό το σημείο συμφωνώ με τον Βέρνερ για αυτό που ε, πρέπει να κάνουμε. Όμως τώρα όσον αφορά τα διαφορετικά επίπεδα, το δικό μας επίπεδο πρέπει να είναι εκείνο του οράματος. Και αν μιλήσουμε για μια αληθινή, πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση, τότε πρέπει να αρχίσουμε με το βαθύ χάσμα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Κάποιες περιοχές στην Ευρώπη έχουν αυξανόμενη φτώχεια και ανεργία και περνάνε βαθιά κρίση προσαρμογής και στην Ανατολική Ευρώπη. Τα ίδια πράγματα και σε άλλες περιοχές. Όπως και στη δική μου χώρα, για παράδειγμα, υπάρχει μεγάλη ισροή κινητού κεφαλαίου που, που μειώνει τα επιτόκια και έχουμε ελάχιστους μηχανισμούς για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή τη διαφοροποίηση. Γι' αυτό λοιπόν η κύρια οικονομική συνεισφορά της Επιτροπής μας στο ζήτημα της αληθινής ένωσης είναι η εξή. Πώς μπορούμε να, κάνουμε, να γεφυρώσουμε αυτές τις διαφορές το γρηγορότερο δυνατόν. Πάντα θα υπάρχουν κρίσεις σε αυτές τις περιοχές, αλλά πρέπει να τις ξεπεράσουμε με μεταρρυθμίσεις σε αυτές τις περιοχές. Αλλά χρειαζόμαστε επίσης και ισχυρότερα εργαλεία. Και στον κατάλογο των εργαλείων αυτών πρέπει, και πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη αναφορά, είναι οι ξεκάθαρες προτάσεις ως προς το πώς να συσταθεί αυτό το όργατο και να περιοριστούν οι διαφοροποιήσεις στα επιτόκια. Επίσης πρέπει να προτείνουμε ισχυρούς αυτόματους σταθεροποιητές, ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη. Οι αυτόματοι σταθεροποιητές τι είναι. Είναι ένας κοινό ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ικανού μεγέθου που θα χρησιμοποιείται για να χρηματοδοτούνται ε, επενδυτικά μέσα αλλά και για να σταθεροποιηθεί οι, κοινωνικοί, οι κοινωνικές συνθήκες στις πιο δύναμες περιοχές έτσι ώστε η προσαρμογή να γίνει πιο γρήγορα. Η πρόταση λοιπόν αυτή που υπερασπίστηκαν πολλοί οικονομολόγοι ε, για το σύστημα Αντιμετώπιση τη ανεργία είναι ένα όραμα το οποίο πρέπει να υπερασπιστεί το Κοινοβούλιο. Συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν για την φορολόγηση. Ε, ασχολούμαστε πάρα πολύ με την φοροδιαφυγή, αλλά πρέπει να, ε, για την ε, φορολογική απάτη, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για τα ελάχιστα πρότυπα στον κοινωνικό χώρο. Τέλος, τελευταία πρόταση, Πρόεδρε, όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο με μια ισχυρή δημοκρατική συζήτηση με του πολίτε. Επομένω, εάν μιλάμε για ένα όραμα ω Κοινοβούλιο, πρέπει επίση να μην ξεχάσουμε και την ε, δημόσια συζήτηση. Δεν μπορούμε να, το, να κάνουμε συζήτηση μόνο εδώ στα όργανα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προλάβαμε να τελειώσουμε. Για όσους δεν βρίσκονται εδώ, το Συμβούλιο της ΕΚΟΦΗΝ, στο Συμβούλιο της ΕΚΟΦΗΝ το τελευταίο Σαββατοκύριακο είπα ότι το Κοινοβούλιο ανέφερε ότι η επίλυση της κρίσης είναι πάρα πολύ σημαντική και το πρώτο βήμα σε αυτό που λέω επίλυση κρίσεων, πέτυχε. Φαίνεται λοιπόν ότι μας ζητείτε να προχωρούμε βήμα-βήμα. Εντάξει, καλό είναι αυτό, μπορούμε. Αυτό που δεν μπορούμε είναι να προχωρούμε προς τα πίσω. Και πραγματικά, όταν αναφερόμαστε σε, στις εποπτικές ε, πτυχές της ε, ΕΚΤ, είναι κάτι που θα γίνει σε άλλο κείμενο. Αλλά θέλω να πω ότι όταν αναφερόμαστε λοιπόν σε αυτό, αν δεν έχουμε τη δομή από πίσω μας, τότε χρειάζεται ένα, να, συσταθεί, να αναφερθούμε σε ένα καινούργιο επίπεδο του ε, αντιμετώπισης με τα εθνικά κοινοβούλια. Γιατί εάν υπάρχει αυτό το, αυτή η ραχοκοκαλιά, τότε τα εθνικά κοινοβούλια θα μπορούν να στηριχτούν σε αυτά. Έτσι, εάν λείπει αυτό, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να προχωρήσουμε μπροστά. Γι' αυτό και συμφωνώ με όσους ανέφεραν ότι πραγματικά πρέπει να ασχοληθούμε με όλους τους πυλώνες ταυτόχρονα. Είναι πιο λογικό. Σίγουρα θα το συζητήσουμε όταν φτάσουμε στον τομέα της εποπτείας. Και οι λεπτομέρειες μπορούν να πάνε στην ε, άλλη έκθεση της Μαριάν και του Σβέν. Στην έκθεση, στη μορφή της έκθεσης, ίσως ε, θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο καινοτόμοι και θα ήθελα να ζητήσω από την Αρμόδια να το παρουσιάσει με κάποια πιο εύπεπτη μορφή. Διότι αυτή που έχουμε τώρα δεν είναι. Υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία λέμε εκτιμώντας ότι κτλ. κτλ. Και πιστεύω πως είναι καλή πολιτική δήλωση να υπάρχει αυτό το εκτιμώντας. Μία επιλογή είναι αυτή. Ας δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε ως Επιτροπή για να βοηθήσουμε την Μαριάν. Αλλά τονίζω, δεν φταίει εκείνη για όλες τις διαφωνίες. Μαριάν, σε πέντε λεπτά δεν θα έχουμε διερμηνία, αλλά αν θέλεις να πεις ε, κάποια τελευταία πράγματα, τώρα είναι η ώρα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είχα αρκετό χρόνο στην αρχή για να παρουσιάσω τα βασικά σημεία αυτής της έκθεσης και να τραβήξω την προσοχή όλων, ούτω ώστε κανένας μετά να εκπλαγεί περαιτέρω. Άκουσα λοιπόν με προσοχή αυτά που είπανε οι συνάδελφοι και όταν θα τα έχουμε όλα πλέον σε χαρτί θα μπορέσουμε να συζητήσουμε καλύτερα. Και θα δούμε πώς ε, θα βρούμε καλύτερες λύσεις. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, ε, τους σκιώδεις εισηγητές, ε, όλους όσους πήραν το λόγο. Διότι Πρέπει να ακούσουμε πρώτα τους συναδέλφους και μετά να φανταστούμε την όλη διάρθρωση του κειμένου. Πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ μακρύ και χρειάζεται να το συντομεύσουμε. Πρέπει να συνεννοηθούμε και με τη γραμματεία την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Θα κοιτάξουμε να δώσουμε μία μορφή στην διάρθρωση της έκθεσης. Πάντως εγώ είμαι σύντομη γενικώ. Δεν μπόρεσα να είμαι όμω πιο σύντομη από αυτό. Διορία για τι τροπολογίε 24 Σεπτεμβρίου. Συζήτηση 8 και 9 Οκτωβρίου για να ψηφίσουμε στις 15 Οκτωβρίου. για να διαβάσουμε γέρο το μήνυμά μας. Επόμενη συνεδρίαση 24 Σεπτεμβρίου, 3 το απόγευμα δημόσια ακρόαση για το διατραπεζικό επιτόκιο Λίμπορ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους διερμηνείς για την ε, μικρή υπέρβαση ωραρίου. Μία ερώτηση. Στις 26 Σεπτεμβρίου είπαμε είναι, αλλά στις 26 Σεπτεμβρίου υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικότερο. Δεν υπάρχει ακρόαση που να είναι επιβεβαιωμένη, διότι ακόμα δεν έχουμε συμφωνήσει γι' αυτό. Έχουμε κάποια άλλη ημερομηνία, εν υπάρξει ε, συμφωνία και αυτό το είπα στην αρχή χθες.